Mes chers collègues, αρχίσουμε λοιπόν την συνεδρίαση. Δεν είναι βέβαια παρόντες ακόμη όλοι παρόντες. Ε, η... Μεγάλος αριθμός μελών του Λαϊκού Κόμματος είναι στο Παλέρμο την εβδομάδα αυτή. Ε, αυτά βέβαια και ορισμένοι σοσιαλιστές λείπουν, ε, διευκολύνουν τις ψηφοφορίες. Έχουμε μια ημερήσια διάταξη που δεν είναι πολύ φορτωμένη, άρα θα προσπαθήσουμε ασφαλώς βέβαια να την διεξέλθουμε με την δέουσα προσοχή αλλά ίσως κατορθώσουμε να τελειώσουμε λίγο νωρίτερα ώστε αμέσως μετά να περάσουμε στην συνεδρίαση των συντονιστών εποφελούμενοι βέβαια έτσι της παρουσίας των μεταφραστών μέχρι τις 12.30. Ένα. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ορισμένες τροποποιήσεις τώρα. Το 9 που προβλέπει την γνωμοδότηση του κυρίου Αμπάντ μετά από δική του ε, αίτηση αναβάλλεται για τις 22-23 ε, Μαΐου. Το 10 και το 11 γνωμοδότηση της Utah Hawk για τους οργανισμούς ΕΝΙΣΑ και ΕΜΣΑ συζητήθηκαν την προηγούμενη Δευτέρα στην συνεδρίαση και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπενθυμίζω ότι μέχρι τις 16 Μαΐου 12 το μεσημέρι ισχύει η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και ψηφοφορία προβλέπεται 15 έκτου. Για το 7 τώρα, για την πράσινη βίβλο του κ. Χαγκλούντ πάλι μετά από έντηση του εισηγητού, σας προτείνω αναβολή για την επόμενη συνεδρίαση. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη γνωμοδότηση Χάγκλουντ, για την οποία ε, θα λάβει το λόγο όταν έρθει η ώρα. Ο κ. Χάγκλουντ είναι παρόν και νεύει καταφατικά στα όσα λέω. Αν δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις. Καλημερίζω και τον κύριο Μπέγκε που είναι βασικός εκπρόσωπος σήμερα του Λαϊκού Κόμματος έχοντας προτιμήσει τις Βρυξέλλες από το Παλέρμο. Άλλο σχόλιο δεν έχω. Εγκρίνεται η σε διάταξη. Για τις ανακοινώσεις τώρα του Προέδρου έχετε το ε, τεύχος κόμπου νιούς και τις γλώσσες που προβλέπονται σήμερα. Επίσης ε, μεταδίδεται από το ίντερνετ η συνεδρίασή μας, το λεγόμενο web streaming. Ας προχωρήσουμε στο θέμα 3 της ημερήσιας διάταξής μας. Αρχίζει δηλαδή η εργασία για το σχέδιο προϋπολισμού 2012 και το σχέδιο εντολής για τον τριμερή διάλογο. Η συγγήτρια κυρία Μπαλζάνη έχει ήδη καταθέσει ένα σχέδιο. Ας λάβει αμέσως τον λόγο για να παρουσιάσει το σχέδιο αυτό. Η Φραντσέσκα λοιπόν έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 20 Απριλίου ο Επίτροπος κύριος Λεβαντόσκι κατέθεσε το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια, η πρόταση αυτή γίνεται σε δύσκολη περίοδο. Η 20 Απριλίου ήταν δύσκολη περίοδος γιατί ήταν μόλις πριν από τις διακοπές δεν υπήρχαν ακόμα πια κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και γι' αυτό μαζί με την γραμματεία, την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερος, χρειάστηκε να εγκύψω στην ε, έκθεση αυτή, αλλά δεν μπόρεσα να συνενωθώ με άλλους συναδέλφους γιατί έλειπαν σε διακοπές. Άρα τώρα επισημαίνω σήμερα ότι πρόκειται για ένα ανοιχτό έγγραφο, ανοιχτό δηλαδή σε όλες τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις των συναδέλφων από τις ε, διάφορες πολιτικές ομάδες, παρεμβάσεις οι οποίες θα είναι σημαντικές για τον εμπλουτισμό του εγγράφου. Πρόκειται για εντολή σε σχέση με μια διαπραγμάτευση. Θα δείτε ότι λείπει το τελεκό μέρος, εκεί δηλαδή όπου καθορίζονται οι διαπραγματευτικές γραμμές. Για το κοινοβούλιο δηλαδή. Ακριβώς αυτό, αυτή η σύνοψη θα ήθελα να ε, συνταχθεί μετά από τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων. Στη διάρκεια της συνταλλαγής απόψεων θα διατυπωθούν και τροπολογίες και βεβαίως η εργασία αυτή θα συνεχιστεί τον Μάιο. Πρόκειται για έγγραφο όπως είπα από την αρχή ανοιχτό σε παρεμβάσεις. Το δε τελικό μέρος, το τελευταίο μέρος θα γίνει αντικείμενο επεξεργασίας με συνοπτική μορφή και εν τέλει θα δίνει την τελική κατεύθυνση για την εντολή. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω προκαταρκτικά. Θα ήθελα τώρα να σας αναπτύξω ορισμένες σκέψεις για τα πιο σημαντικά σημεία. Αυτό που θα ήθελα οπωσδήποτε να υπογραμμίσω και που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Κομισιόν τόνισε ιδιαίτερα τη συμβολή που κάνει η πρότασή της στη 2020 δείχνοντας έτσι πως θέλει να δεχθεί το αίτημά μας του να ξεκινήσουμε και να οικοδομούμε μια πορεία προς την επίτευξη της στρατηγικής 2020. Το 43,5% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα χρηματοδοτήσει τις ε, γραμμές της στρατηγικής 2020. Ωστόσο θα πρέπει να βασιστούμε στη διαφάνεια γιατί ένας αριθμός μόνος του δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν πως όταν υποδείξαμε τις κατευθυντήρες γραμμές για το 2012, ως Κοινοβούλιο γενικά δεν επικαλεστήκαμε, ούτε υπενθυμίσαμε τη στρατηγική 2020, αλλά ε, εντοπίσαμε κάποιους στόχους της στρατηγικής αυτής απασχόληση, ανάπτυξη, έρευνα και ανάπτυξη, ε, καινοτομία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες πράσινες τεχνολογίες. Προς αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση λοιπόν θα πρέπει να μετρήσουμε συζητήσουμε ουσιαστικά τη συμβολή του προπολογισμού στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 2020. Κυρίως όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα των αυξήσεων και είναι αρκετά εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο όσον αφορά τον τίτλο 3, την κατηγορία 3α, αφορά όχι αυξήσεις στρατηγικής σημασίας που είναι οι θελημένες πολιτικός, αλλά είναι αυξήσεις που είναι φυσιολογικές και ήδη είχαν αποφασιστεί στην αρχή της, ε, του δημοσιονομικού προγραμματισμού ε, για το 2007 μέχρι το 2013 και αυτό μας ε, υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε αυτές τις επιλογές. <clears throat> Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε δηλαδή πού θέλουμε να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα στρατηγικής σημασίας, πέρα δηλαδή από την αρχικό προγραμματισμό που είχαμε ορίσει για την περίοδο 2007 με 2013. Κάτι ακόμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ο πληθωρισμός. 2,7% που τοποθετεί σε νέες διαστάσεις πολύ έντονα το επίπεδο των υποχρεώσεων και των πληρωμών. Η αύξηση 3,7% των υποχρεώσεων με βάση τον πληθωρισμό 2,7 καταλήγει σε ένα απλό 1% και κυρίως το επίπεδο των πληρωμών το 4,9% μειώνεται στο 2,2% δηλαδή είναι μια μεγάλη μάλλον μοιράζουμε στη μέση το ποσοστό του, του πληθωρισμού. Το 80% του πληθωρισμού είναι η συνδιαχείριση των κρατών μελών. Οι πληρωμές δεν είναι μόνο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά είναι ένας τρόπος για να μειώσουμε ε, ας πούμε και την ε, προσβασιμότητα στα έγγραφα τα οποία θέλουμε να εξετάσουμε. Βασιζόμαστε λοιπόν σε εκτιμήσει των κρατών για να ορίσουμε το επίπεδο των πληρωμών και θα έλεγα ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα να μην δεχτούμε καμία μείωση. Για να μην επηρεάσουμε την ίδια την υλοποίηση, την εκτέλεση μάλλον του προϋπολογισμού. Πάντοτε τώρα σε σχέση με την ε, νέα ερμηνεία, μάλλον την ε, ερμηνεία του κανονισμού, του προϋπολογισμού, συγγνώμη, όχι μόνο ω προπολογισμό του 2012, αλλά σε συνδυασμό με ολόκληρο το δημοσιονομικό πανόραμα και εικόνα ε, αυτό προσπαθώ να εκφράσω στις παραγράφους 16, 17 και 18. Γιατί Εάν δούμε δεδηλωμένε αυξήσει και τις τοποθετήσουμε μέσα σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο που σας λέω, θα δούμε ότι πολλές γραμμές του προπολογισμού που είναι πολύ σημαντικές για τη στρατηγική 2020, όπως το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, όπως το Progress, το Μαρκοπόλο, το Γαλιλαίο, αυτά τα προγράμματα μειώνονται ως κονδύλια μέχρι το 2013 ενώ άλλα όπως ε, τα ευρωπαϊκά δίκτυα, τα, τα δίκτυα για την ενέργεια, το έρασμος κτλ αυξάνονται με πολύ πιο τρόπο. Δεν φτάνουν ούτε στην αύξηση του 5% που επιτρέπεται με βάση το άρθρο 37 της Διοργανικής Συμφωνίας και κυρίως μέγα τμήμα της αύξησης που δηλώνει η Κομισιόν για την κατηγορία 1 στις υποχρεώσεις 12,6% και στις πληρωμές 8% καθορίζεται από, με μαθηματικό τρόπο από τις από τα 750 εκατομμύρια που έχουν ε, ήδη ε, θεωρηθεί δεδομένα, ενώ η συμφωνία δεν υπάρχει ακόμα για το ίτερ προστίθενται ωστόσο άλλα 64 εκατομμύρια περικοπών. Και αυτά είναι πολύ βεβαίστα από πολιτικής άποψης, γιατί μαζί με τον αθλητισμό και τον χώρο της ενέργειας, μια νέα αρμοδιότητα της συνθήκης της Λαβώνας και μια από τις αρμοδιότητες επί των οποίων εμείς πρέπει να παρέμβουμε και να κερδίσουμε όσο γίνεται περισσότερο, Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να μπουν περισσότεροι πόροι για την ε, έρευνα όσον αφορά την ανεξαρτησία μας, την επάρκεια, τη βιωσιμότητα των ενεργειακών μας προγραμμάτων. Έχουμε έπειτα τις γραμμές ε, στην κατηγορία 3α που αφορούν την μετανάστευση. Τρία από τα τέσσερα προγράμματα αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό, αλλά όχι για κάποια επιλογή που συνδέεται με τις επίγουσες ανάγκες, αλλά για αυτήν που ήταν αρχικά η δημοσιονομική ε, πρόβλεψη για την περίοδο 2007-2013. Δεν αυξάνεται καθόλου το κονδύλι για τους πρόσφυγες, πράγμα που θα ήταν χρήσιμο για να ανταποκριθούμε στην επίγουσα κατάσταση στη Μεσόγειο, πράγμα το οποίο καθιστά προφανές και αυτό που θα είναι η χρηματοδότηση του Frontex. Όπως έλεγα και πριν στην κατηγορία 3β, δυστυχώς δεν προβλέπονται <clears throat> γραμμές για τη χρηματοδότηση του αθλητισμού που είναι στην αρμοδιότητά μας και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ενώ στην κατηγορία 4 υπογραμμίζω ότι ο διπλασιασμός του διαθέσιμου περιθωρίου σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά καθοριστεί μέσω των δημοσιονομικών προπτικών συνδέεται με τον κίνδυνο ότι πρόκειται για εξοικονομήσεις που γίνονται από άλλα σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Ε, πολύ σημαντικά προβλήματα γιατί οι νέες προκλήσεις ας πούμε για τη δημοκρατία ως ολόκληρη τη Μεσόγειο ε, δείχνουν ότι ε, πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από τώρα ε, αυτή την κατάσταση και κυρίως τον επόμενο χρόνο. στην κατηγορία 5, πέρα από τον προγραμματισμό που είχαμε δηλώσει την περασμένη χρονιά, ότι δηλαδή θα πρέπει να προσέχουμε οι εξοικονομήσεις να μην καθιστούν δύσκολη τη λειτουργικότητα των προγραμμάτων μας. Δηλαδή να είναι εξοικονομήσεις που εμφανώς συνδέονται με τις διοικητικές δαπάνες, αλλά στην πράξη μετά μπορεί να αποδειχθεί ότι πρόκειται για περικοπές στη λειτουργικότητα και στην απόδοση των προγραμμάτων. Αυτό το έχω ήδη εδώ βάλει γιατί είχε προκύψει στην πρώτη συζήτηση που είχαμε στις 20 Απριλίου και ζητώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Και επίσης να προστατευτεί η διαφάνεια, να είμαστε βέβαιοι ότι σε μια φάση λιτότητα, ναι, είναι σημαντικό να κάνουμε εξοικονομήσει, αλλά όχι να βλάψουμε ε, εργαλεία ή μέσα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και που μπορεί να αποδειχθούν μια χαμένη ευκαιρία που θα μπορούσε αντίθετα να δώσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Φραντσέσκα για την γραπτή έκθεση και για την πολύ σαφή προφορική παρουσίαση. Ο κύριος Μπόκρος είναι ο πρώτος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω σημαντικά προβλήματα με την έκθεση επί της ουσίας, σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, αλλά και από πλευράς τακτικής. Ας ξεκινήσω από το θέμα της στρατηγικής, όχι στατιστικής στρατηγικής. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι από πλευράς Κομισιόν αποτελεί σημαντικό επίτευγμα το ότι προτείνουν ε, αύξηση κατά 4,9% για του χρόνου, συνολικά για τον προϋπολογισμό. Συμφωνώ απόλυτα με πολλά από όσα ανέφερε η Φραντσέσκα. Δηλαδή, και οι πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και οι οικονομικές προτεραιότητες, κυρίως από πλευράς Κομισιών, δεν σημαίνει ότι ανταποκρίνονται κατά ανάγκη ναι, σωστά και στα νούμερα και στη δομή του προϋπολογισμού στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι σε κάθε περίπτωση θα λέμε ότι λυπούμεθα που δεν υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση. Και όλο το έγγραφο αυτό κάνει. Όλο λυπάται, όλο εκφράζει τη λύπη του. Τουλάχιστον σε 30 περιπτώσει. Ε, λέγεται πολύ ξεκάθαρα ότι λυπούμεθα που δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη ή αύξηση και δεν υπάρχει ούτε μία πρόταση που να λέει περισσότερη μείωση. Α κάνουμε περί μεγαλύτερη μείωση. Α ε, το πάρουμε απόφαση. Μακάρι το Δεκέμβριο να υπάρχει αύξηση 4,9% αλλά δεν νομίζω να υπάρχει. Μέχρι το Δεκέμβριο σας διαβεβαιώ ότι και 3% να είναι θα μας ικανοποιήσει πάρα πολύ. Γιατί αυτό έχει κατά νου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά και ίσως και λιγότερο, αν κανείς ρωτήσει ορισμένε από τις κυβερνήσεις. Ας δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιχειρήματα, σε πολλές περιπτώσεις αυτά δεν είναι συνεπή. Ας δούμε το σημείο 5. Το να λέμε στο σημείο 5 ότι δεν έχει νόημα να μειωθεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με το συνολικό τεράστιο εθνικό χρέο των 27 κρατών μελών. Πραγματικά αυτό δεν είναι συνεπές και δεν υπάρχει καμία σχέση. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και συνετοί στον προπολογισμό. Όχι λόγω του μικρού μεγέθους, αλλά γιατί θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στους φορολογούμενους, στους οποίους και λογοδοτούμε και πρέπει να δαπανούμε τα χρήματά τους ε, σωστά και υπεύθυνα. Άρα δεν πρέπει να κάνουμε μείωση επειδή είναι πολύ μικρός προβλήμα σε σχέση με το χρέος. Αυτό είναι ένα κακό επιχείρημα. Γιατί ακριβώς περί του αντιθέτου πρόκειται. Όταν υπάρχει ένα τόσο τεράστιο χρέος στους εθνικούς προπολογισμούς ε, και στο δημόσιο τομέα των κρατών μελών, έχουμε ακόμη ένα λόγο να είμαστε πιο συνετοί και να ελέγχουμε όλα τα κονδύλια του προπολογισμού ένα προς ένα. Και όπως είπε και η Φραντσέσκα, ναι, να προτείνουμε αυξήσει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όπως ε, ε, επισήμανα να προτείνουμε ορισμένες φορές και μειώσεις. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο όμως. Και κάτι τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό η τακτική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Εάν λάβατε υπόψη τα διδάγματα που αντλήσαμε από τις διαπραγματεύσεις της περσινές για τον προπολογισμό και τα θυμόμαστε όλοι, θυμόμαστε πόσο δύσκολο ήταν, για να μην πω τραγικό, κάποιες φορές εξελίξασαν τραγικές, ε, βέβαια με κάθε σεβασμό προς όλους ε, και προς τη Βελική Προεδρία. Δεν νομίζω όμως ότι τα πράγματα θα είναι ευκολότερα φέτος. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάθε συμφέρον να έχουμε με το πλευρό μας την Κομισιόν και να μην είναι με το μέρος του Συμβουλίου. Αλλά νομίζω ότι θα απομακρυνθεί παρά θα πλησιάσει σε εμά η Κομισιόν με αυτό το έγγραφο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Φραντσέσκα Μπαλτσάνη για την πολύ επικοδομητική έκθεση ε, που είναι αυστηρή και εύστοχη. Σε ό,τι τον κύριο Μπόκρος, ας δούμε λίγο την πραγματικότητα. Τι γίνεται επί σειρά ετών. Ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση ως αναλογία προς την ευρωπαϊκή οικονομία μειώνεται. Παρά το γεγονός ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη έχουν επιβάλει ένα σωρό νέους φόρους και νέα προγράμματα στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μπόκρος έδωσε μια πραγματική εικόνα της κατάστασης. Θα έλεγα αντίθετα ότι έχουμε στριμώξει νέες πολιτικές ε, κάτω από την ίδια οροφή, κάτω από την ίδια στέγη και έτσι είχαμε μειώσει πολλούς τομείς. Άρα δεν νομίζω ότι η εικόνα του κύριου Μπόκρος είναι η σωστή αλλά θα πρέπει ε, όταν έρθουμε σε επαφή και με το Συμβούλιο να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Η Κομισιόν νομίζω ότι έχει ακολουθήσει μια πάρα πολύ προσεκτική προσέγγιση προτείνοντας την αύξηση του 4,1%. Αλλά τελικά έχουμε ήδη λάβει πολιτικές αποφάσεις ε, για διάφορα προγράμματα και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να μας είχε οδηγήσει να κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς τα παραπέρα γιατί έχουμε δεσμεύσεις απέναντι και σε περιφέρειες, ε, στις τοπικές αρχές και σε άλλους πολύ σημαντικούς τομείς της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα περιορισμοί, περικοπές μεγαλύτερες από αυτά προτείνει η Κομισιόν δεν θα είναι ευεργετικό για τα κράτη-μέλη όπως λέει ο κύριος Μπόκρος. Θα είναι ευεργετικές οι περικοπές μόνο για κάποια κράτη-μέλη αλλά τα περισσότερα θα πληγούν από τις μειώσεις αυτές. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των δαπανών σε κάποια ε, κονδύλια. Αυτό είναι γεγονός, αλλά αυτό το οποίο εμείς πληρώνουμε ουσιαστικά συνεισφέρει στην ανάκαμψη μετά την κρίση και νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό επιχείρημα της Φραντσέσκα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο ώστε να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Τι θέλουν να κάνουμε εμεί. Έχουν προσθέσει καθήκοντα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στόχοι 2020, το σχέδιο τη Συνθήκης Λισαβόνα, Τι θέλουν να κάνουμε εμεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια στρατηγική συζήτηση για τι προτεραιότητε και ειδικότερα για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάκαμψη. Νομίζω ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό και επικοδομητικό ρόλο και εκεί πάνω θα πρέπει να ε, χαράξουμε τη στρατηγική μας. Αυτό πάντως με ανησυχεί εμένα είναι η κατηγορία 4. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν νέε ανάγκε, ιδίω ό,τι αφορά την πολιτική γειτονία και κυρίω στη Μεσόγειο, στο Νότο. Ε, δεν ξέρουμε ακριβώ ε, ποιε θα είναι οι νέε προτάσεις, νέες ε, ανακοινώσει και η νέα τροποποιητική επιστολή, τη διορθωτική επιστολή της Κομισιόν, αλλά προτείνεται να χρηματοδοτήσουμε κάποιες από αυτές τις προτεραιότητες μειώνοντας κάποια προγράμματα αναπτυξιακά, το μέσο DCI κτλ. Δεν συμφωνώ γιατί θεωρώ ότι αυτά είναι προτεραιότητες σημαντικές για μας από πολιτικής πλευράς και δεν είναι ε, ο σωστός τρόπος να περικόπτουμε τις δυνατότητες που έχουμε για να συνεισφέρουμε στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας ή στο να ε, συνεισφέρουμε στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρηματοδοτήσουμε τις νέες προτεραιότητες στη Μεσόγειο. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε αυτό που ε, χρησιμοποιούν ως δικαιολογία, ως επιχείρημα είναι ότι τουλάχιστον εν μέρη η χαμηλή εφαρμογή είναι ένα πρόβλημα, παραδείγματο χάρη με το πρόγραμμα ΙΠΑ. Αλλά αυτό δεν είναι λόγο να γίνουν περικοπέ, γιατί μιλάμε για πολιτικέ προτεραιότητε. Άρα να βελτιώσουμε την εφαρμογή, την υλοποίηση. Αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα και πρέπει να το προσπαθήσουμε. Και κάτι άλλο που με ανησυχεί είναι κάποιε από τι περικοπέ στην κατηγορία 5. Διότι αν περικόψουν τι διοικητικέ δαπάνε πάρα πολύ, τότε δεν έχουμε και πάρα πολλέ δυνατότητε και μέσα να βελτιώσουμε την υλοποίηση, γιατί χρειαζόμαστε και προσωπικό για αυτό το λόγο. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ναι, μεν μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί, αλλά πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου τις προτεραιότητές μας και να μην ε, χρηματοδοτήσουμε τη Μεσόγειο κοντόθωρα, μειώνοντας ε, τα προγράμματα της ΕΑ και ΕΙΠΑ. Είναι πολύ καλή έκθεση της Φραντσέσκα. Τώρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προσθεθούν στο τέλος κάποιες παράγραφοι γιατί είναι διτός ο στόχος της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα, γενικά να ε, κάνει κάποιες σκέψεις για το σχέδιο προπολογισμού και να ε, ο, ιεραρχήσει κάποιες προτεραιότητες, αλλά δεύτερο είναι η εντολή για τον τριμερή διάλογο. Και πρέπει να δούμε. Μπορούμε τελικά να πετύχουμε κάτι σε αυτόν τον τριμερή διάλογο. Μέχρι στιγμής ε, ε, δεν είχαμε επικοδομητικό τριμερή διάλογο. Τον Ιούλιο όχι, δεν τα καταφέρνουμε. Πριν από 10 χρόνια, ναι, όταν ήμουν συγκητής το 2003 που είχαμε λύσει τον Ιούλιο τότε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά αυτό ήταν μία φορά. Άπαξ έγινε. Ας προσπαθήσουμε αυτή τη φορά τουλάχιστον κάποια πράγματα να τα διευθετήσουμε. Κάπου να καταλήξουμε τέλος πάντων κατά τον τριμέρι διάλογο του Ιούλιο Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ να λέει ο πρόεδρο. Άρα αυτό που συγκρατούμε είναι ότι στόχο μα αυτή τη φορά είναι να είμαστε αποτελεσματικοί στον ε, τριμερή διάλογο όσο είμαστε χάρη στον τότε εισηγητή μα το 2003. Ωραία. Πολύ καλά. Χάγκλουντ για του φιλελευθέρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όλοι θέλουμε να αποφύγουμε την κατάληξη την περσινή το Δεκέμβριο και από αυτή την άποψη Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το τι λέμε και τι βάζουμε σε αυτά τα έγγραφα. Εν γέννη πιστεύω ότι το μεγαλύτερο τμήμα του εγγράφου, όπως το παρουσιάζει η συγγήτρια, είναι καλό και θέλω να την ευχαριστήσω γι' αυτό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σκεφτούμε τι επιδιώκουμε. Πάντοτε έχοντας υπόψη μας την κατάσταση πέρσι το Δεκέμβριο. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στα όσα επιδιώκει η συγκήτρια και ο κύριος Μπούκρος. Γιατί αν δεν τα καταφέρουμε και με βάση τις αντιδράσεις κάποιων κρατών μελών ε, στην πρόταση της Κομισιόν πριν το, Πάσχο, πριν το Πάσχα, δεν φαίνεται να είναι εύκολη η κατάσταση. Και πρέπει να το αποφύγουμε, επαναλαμβάνω, λαμβάνοντα υπόψη ότι, ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είπατε για το 2,7%. Μιλάτε για εκτίμηση της Eurostat. Πού βασιστήκατε για αυτά τα στοιχεία. Γιατί αν δεν είναι σωστά επηρεάζουν πάρα πολύ ολόκληρη, την, ολόκληρη το, το, το σχέδιο. Εγώ προσωπικά καλωσορίζω το γεγονός ότι και η Κομισιόν προσπάθησε να αναζητήσει αρνητικές προτεραιότητες είναι με ένα αρνητικό όρο. Μιλάμε για ανακατανομή και είναι μια πολύ φυσιολογική διαδικασία στον δημοσιονομικό προγραμματισμό. Πρώτα ψάχνεις να δει που μπορεί να ανακατανείμεις ποσά και μετά ζητά παραπάνω χρήματα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει και εμείς να μπορούμε να το κάνουμε αυτό και η Κομισιόν αυτό έχει κάνει. Και αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να την καλωσορίσουμε. Από όσα κατάλαβα από είπε ο Γιώραν, Φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες τέτοιες ανακατανομές τις οποίες δεν ε, θα ήθελαν κάποιες ομάδες, αυτό το κατανοώ, αλλά ως ε, ιδέα δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κατά της ανακατανομής των κονδυλίων. Είναι καλή εξέλιξη αυτή. Τώρα για την ευελιξία. Φραντζέσκα, έχουμε καθόλου αριθμούς για ολόκληρο το εμ, σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Πόσο, σε τι αντιστοιχεί το 5% αυτό. Θα ήταν σημαντικό να έχουμε αυτή την ενημέρωση πριν μπούμε στις διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η δεύτερη μου ερώτηση. Και έπειτα μια σύντομη παρατήρηση, στην οποία θα πρέπει να επανέλθω όταν θα εξετάσουμε τη δική μου γνωμοδότηση που θα σας παρουσιάσω, το πρόβλημα ITER. Twitter. Πριν από λίγες εβδομάδες, όταν μας παρουσίασε η Κομισιόν το σχέδιο προπολογισμού της για τον επόμενο χρόνο, αν δούμε το ποσό που χορηγείται στην έρευνα, όταν το δει κανεί από πρώτη ματιά φαίνεται πολύ καλό. Αλλά αν αφαιρέσει κανεί τα χρήματα που είναι μόνο για τη χρηματοδότηση των προβλημάτων Twitter, δεν μένει φράγκο για την υπόλοιπη έρευνα. Η αύξηση δηλαδή είναι στο, στο χαρτί μόνο και αφορά το ίτερ. Το ίτερ όμως είναι πολύ αμφισβητήσιμο. Και δεν είμαι λοιπόν ευχαριστημένος γι' αυτό. Θα επανέλθω στην ε, γνωμοδότησή μου όταν θα σα την παρουσιάσω για αυτό το θέμα. Αλλά θα ήταν καλό το έγγραφο τούτο εδώ να είναι σύμφωνο με τη δική μου γνωμοδότηση για τι ρυθμίσει τη Βρατόμα. Ε, το σημείο λοιπόν 20 εδώ που μιλά για το ίτερ ε, στην κατηγορία 1α θα ήταν καλό να συμφωνεί. Πολλά χρήματα λοιπόν θα επιστραφούν στα κράτη-μέλη γιατί ε, ε, δεν χρησιμοποιήθηκαν το περασμένο χρόνο. Τεράστια ποσά και έτσι αυθόρμητα θα έλεγα ότι αυτά τα χρήματα, αν και ξέρω πως υπάρχουν τεχνικά καλές εξηγήσεις για το ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθούν τα προβλήματα του ίτερ, από πολιτικής άποψης όμως τα χρήματα αυτά καλύτερα θα ήταν να χρησιμοποιηθούν εδώ ε, για το ίτερ και να μην τρώνε σαν τους κανίβαλους το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Για το ίτερ λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση ότι, που είναι αμφισβητήσιμη, είναι και πολύ κακό δημοσιονομικό προγραμματισμό. Η Κομισιόν δεν έλαβε υπόψη ότι επανειλημμένω είπαμε πω δεν δεχόμαστε τη λύση ίτερ. Και μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει καμιά αλλαγή στο προγράμματα τη Κομισιόν για τη χρηματοδότηση του ίτερ. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο λοιπόν με αυτό το θέμα. Αυτό βέβαια δεν αφορά την ίδια την έκθεση, αλλά το ίτερ. Εν γέννη πάντως, νομίζω πως μπορούμε να βρούμε μια κοινή βάση εδώ με μικρές προσαρμογές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ανδρέασεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης και την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Στηρίζω τα σχόλια του κ. Μπόκρος και δεν θα τα επαναλάβω. Η προσδοκία του για 3% αύξηση εξακολουθεί να είναι υψηλή. Αυτό θα πω μόνο. Λίγα σχόλια. Πρώτο, ουδής χαίρεται για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα λεγόμενα ραλ, τα υπόλοιπα δηλαδή, τα ρευτοποιήσιμα υπόλοιπα. Δεν εντάσσονται στις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει δείχνουν όμως ότι οι χώρες μέλη δεν μπορούν να απορροφήσουν τα προγράμματα για τα οποία έχουν δεσμευτεί. Αυτό θα είναι και το πρώτο θέμα, θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα που συζητούμε όταν συζητούμε τον προπολογισμό. Και νομίζω ότι αυτό έχει και στρεβλωθεί και ε, παραγνωριστεί. Και μάλιστα ε, πάρα πολύ σημαντικά. Δεύτερο, η έκθεση απέχει από την πραγματικότητα. Θα έρθω στην παράγραφο 53. Πώς μπορεί να επικρίνει η εισηγήτρια το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφάσισε να μην περιλάβει προγράμματα σχετικά με τον αθλητισμό. Λοιπόν πολύ, αλλά ο αθλητισμός σε περίοδους κρίσεως δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας αυτό το παράδειγμα ως αφετηρία, θεωρώ ότι η συνολική αυτή παρουσίαση του προπολογισμού είναι εκτός πραγματικότητας. Ευχαριστώ κύριε Τρίπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Φραντσέσκα για την εργασία της. Η εκτίμησή της είναι ότι το προτινόμενο επίπεδο ε, από τον Επίτροπο είναι 4,9% συν και ότι είναι το απολύτω απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν υποχρεώσει που έχουν αναλυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Θα τονίσω, γνωρίζω βέβαια ότι υπάρχει εδώ σύγκρουση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων, ορισμένοι θεωρώ ότι είναι πολύ υψηλό ήδη, αλλά γνωρίζουμε και τον Λεβαντόφσκι και γνωρίζουμε ότι είναι άνθρωπο πολύ προσεκτικό σε ό,τι αφορά την αύξηση του προπολογισμού. και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι οι επίτροποι συλλογικά έχουν αντιληφθεί ότι εάν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε όσα θα έπρεπε να κάνουμε, διότι αυτό, αυτά εγκρίθηκαν μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, τότε χρειάζονται τα χρήματα, τα ποσά αυτά. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να είναι να συμπαραταχθεί με το Συμβούλιο, δηλαδή 3% ή και λιγότερα, όπως είπε η κυρία Αντρέασεν, ρόλος δικός μας θα πρέπει να είναι να προβάλλουμε περισσότερο το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον με τις πολιτικές που έχουμε εγκρίνει. Και επομένως εδώ υποστηρίζω την Φρανσέσκα καθώς και τις άλλες πολιτικές ομάδες που πιστεύουν τα ίδια. Θα είναι λάθος να επανέλθουμε τώρα στρατηγικό στην θέση του Συμβουλίου διότι τότε παρετούμεθα από κάθε υποστήριξη της πολιτικής μας. Ενώ αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Γνωρίζω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι αν παρετηθούμε τώρα από την προσπάθεια αυτή θα είναι στρατηγικό σφάλμα. Όταν θα έλθουμε τώρα, θα έλθουμε μάλλον τώρα στις προτεραιότητες, ως μέλος της ομάδας των πράσινων θα πω ότι δεν υποστηρίζω το επίπεδο των πληρωμών, εάν δεν κατευθύνονται αυτές σε ορισμένους στόχους και κυρίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα, οικονομική μεταρρύθμιση και κοινωνική συμπερίληψη. Αυτό σημαίνει ότι θα δεχθούμε εμείς περικοπές όταν αυτές δίνονται σε εσφαλμένους στόχους, ε, τα ποσά δηλαδή δίνονται σε εσφαλμένους στόχους κατά τη γνώμη μας, για παράδειγμα στη Γεωργία, αλλά βεβαίως θα θέλαμε να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια αυτά για να στηρίξουν πιο βιώσιμες πολιτικές. Συνολικά εκτιμώντας τις προτάσεις της Φρανσέσκα, θεωρώ ότι έχει περιλάβει πολλούς θετικούς στόχους και της Ευρώπης 2020 και ορισμένες από αυτές τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητε για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, πρόθεση ανανεώσιμων ενεργειών. Ορισμένες από τις προσεγγίσεις αυτές βλέπω να λείπουν στην κατηγορία 1β, ίσως πρέπει να ενισχυθούν. Τώρα βέβαια θα έρθω και στα σημεία κριτικής, διότι λυπούμε ιδιαίτερα και εδώ συμπαρατάσσομαι λίγο με τον Καρλ Χάγκλοντ, η απόλυτη έλλειψη κριτικής της φιλοπυρηνικής ε, προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μας, για μένα είναι πολιτικό σφάλμα είναι μια προσέγγιση που στερείται ισορροπίας και τώρα μάλιστα υπέρ του ΙΤΕΡ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περικόπτει και άλλες δαπάνες για την πυρηνική έρευνα. Και αυτό είναι λάθος. Εδώ θεωρώ λοιπόν ότι οφείλει να ασκηθεί κριτική στην έκθεση της ε, Φραντσέσκα, αλλά συνολικά ε, την υποστηρίζουμε την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Τρίπελ. Τέρικ Βόγαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την έκθεση της εισηγήτριας. Νομίζω ότι είναι δύσκολη η δουλειά της να συντάξει την έκθεση αυτή υπό τόσο δύσκολες ε, δημοσιονομικές συνθήκες. Γνωρίζουμε ότι προτείνεται αύξηση από την Κομισιόν, αλλά γνωρίζουμε ότι πολλά κράτη-μέλη στο Συμβούλιο θα επικεντρωθούν κυρίως ή μόνο ε, εκεί που γίνεται λόγος για αυξήσεις. Έχουμε αντιδράσει από κάποια κράτη-μέλη. Θα ζητηθεί σίγουρα πάγωμα Άλλοι μπορεί να μιλήσουν για αύξηση του πληθωρισμού 2,7% αλλά πολύ λίγοι θα δεχτούν το 4,9% τον Ιούλιο στον τριμερή διάλογο. Άρα τι τακτική πρέπει εμείς ως Κοινοβούλιο να ακολουθήσουμε και ως Επιτροπή Προπολογισμών, πόσο σκληρά θα αγωνιστούμε για το 4,9% και αν αγωνιστούμε πώς. Ποια όπλα, ποια εργαλεία έχουμε στο πλαστάσιό μας. Αν θέλουμε επίσης να δεχθούμε περικοπές, ποιες θα δεχθούμε. Θα πούμε στην Κομισιόν παραδείγματο χάρη να γίνουν γενικώ περικοπές παντού ή να, όπως έγινε πέρυσι να πούμε ότι θα πρέπει ε, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε κάποιες προτεραιότητες και να μειώσουμε τους πόρους για σχέδια ή έργα που είναι λιγότερο σημαντικά για το μέλλον. Εγώ νομίζω ότι το σημαντικό είναι να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Να μην κάνουμε περικοπές παντού γιατί υπάρχουν πιο σημαντικά προγράμματα, πιο σημαντικές προτεραιότητες σε σχέση με κάποιες άλλες και αυτή νομίζω θα πρέπει να είναι τακτική μας. Όπω είπαν και άλλοι προλαλήσαντε, παραλαμβάνω πρέπει να δούμε τι προτεραιότητε. Και εγώ ανησυχώ για κάποιε από τι προτάσει τη Κομισιόν. Για παράδειγμα, η Κομισιόν για μια ακόμη φορά προτείνει μείωση 100 εκατομμυρίων ευρώ για την Παλαιστίνη, όπω και κάνει και πέρσι. Τεράστιο σφάλμα κατά την άποψή μου. Τώρα που βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόοδος μετά την συμφιλίωση Φατάχ και Χαμάς, αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε τώρα θα ήταν να υποστηρίζουμε την ειρηνευτική διαδικασία και όχι να μειώνουμε 100 εκατομμύρια το προπολογισμό μα για το κονδύλι αυτό. Είναι λάθο τη Κομισιόν. Επίση, να μην βάζει ε, κονδύλια και στον τομέα του αθλητισμού, γιατί είμαστε ε, φίλαθλοι υποστηρίζουμε τον αθλητισμό, ε, ωφελεί τον κόσμο υπό πολλούς και διαφόρους τρόπους. Άρα πρέπει να χρηματοδοτούμε αθλητικά ε, προγράμματα. Έχει χρηματοδοτήσει κάποια πολιτικά σχέδια η Κομισιόν, αλλά τώρα ε, τελειώνει η χρηματοδότηση και δεν αντικαθίσταται. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να φρούμε χρηματοδότηση και αυτά τα προγράμματα. Πάντως, ως Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνολική στρατηγική, να συζητήσουμε τις προτεραιότητές μας αλλά και την τακτική που θα ακολουθήσουμε προχωρήσουμε στη συζητήση, στον τριμερή διάλογο και στις μελλοντικές συνεδριάσεις της συνδιαλλαγής. Ευχαριστώ, ο James Ellis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρία σημεία θέλω να φέρω. Πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο δεν ακούω στη συζήτηση είναι ποια είναι τα οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ΣΥΠΑ κτλ. Δείτε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ σήμερα με τρισεκατομμύρια εκατομμύρια και με το χρέος ε, πρέπει να αυξηθεί η οροφή του χρέους ε, έχουμε τους, ε, του κόμματο του τσαγιού και του, του του τσαγιού που θα πιέσουν κτλ. Εδώ βλέπουμε σε κάποια κράτη-μέλη τεράστια επίπεδα χρέους ενώ οι Κινέζοι παίρνουν ευρωομόλογα για να χρηματοδοτήσουν τις την οικονομία τους. Τι θέλουμε να κάνουμε γενικά μιλώντας. Στρατηγική 2020. Θέλουμε οι Κινέζοι να χρηματοδοτήσουν το μεγαλύτερο μέρο του χρέου μα ή όλο το χρέο μα, ή θέλουμε να το ξεφορτωθούμε αυτό το χρέο και να δούμε πώ μπορούμε να εξηγιάνουμε τα οικονομικά μα. Και βέβαια αυτό ε, δεν μπορεί να αφορά μόνο του εθνικού προβλήματο και αυτόν ευρωπαϊκό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιε είναι οι αναλήψει υποχρεώσεων που έχουμε. Υπάρχουν κάποιε αναλήψει υποχρεώσεων στα κράτη-μέλη, αλλά επειδή δεν υπάρχουν πόροι, τι κόβουν αυτέ τι ε, δεσμεύσει, αυτέ τι αναλήψει υποχρεώσεων. Όταν λοιπόν έχουν πολύ σωστά κάποιε αναλήψει υποχρεώσεων και βλέπουμε, μα είπε και η Φραντσέσκα πολύ καλά, ε, σε ποιε κατηγορίε πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε και να τι φέρουμε σε πέρα. Έχουμε όμω του πόρου για τι δεσμεύσει αυτέ, για να τι υλοποιήσουμε. Γι' αυτό η πρώτη φορά για πρώτη φορά βλέπω να προτείνει σε κάποιε θέσει ε, και κάποια κονδύλια κομισιών περικοπέ. και αυτό μετά δεν έχουμε πόρου. Δεύτερον, πώ θα προχωρήσουμε. Αυτό που δεν βλέπω είναι έγγραφα εργασία για μεγάλα θέματα, για να μα βοηθήσουν εμά του βουλευτέ που είμαστε μέλη τη Επιτροπή Προκλεισμού να καταλάβουμε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο έγγραφα και έρχομαι σε αυτό που είπε ο Γκόραν Φέρμ. Ποιε είναι οι στατικέ μα προτεραιότητε όλα τα έχουμε ως προτεραιότητες, είπε και ο κύριος Μπόκρος διάφορα. Έχουμε πρόοδο, ναι, αλλά πρέπει να πούμε ποια είναι αυτά που θέλουμε να κάνουμε ως κοινοβούλιο και σε ποια πρέπει να επανέλθουμε, ίσως αργότερα. Τα τελευταία χρόνια στην Επιτροπή μας νομίζω ότι απλά ε, έχουμε δεχθεί και ακούμε τις διάφορες προτεραιότητες, τις βάζουμε όλες στο ίδιο. Καλά, θέλω. Ε, η δουλειά μας ποια είναι. Να πούμε, κοιτάξτε, έχουμε αυτά τα χρήματα και αυτές τις προτεραιότητες προτείνουμε να υλοποιηθούν. Δηλαδή, νομίζω ότι η συζήτησή μας θα πρέπει να αναβαθμιστεί για να συζητήσουμε το προορισμό μέχρι το 2020. Γιατί κάποιες συζητήσεις μας ε, οδήγησαν σε σύγχυση όπως πέρυσι. Θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας για τον προβλησμό του 2020, να δούμε πού θα πάει ο υπολογισμός, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες, πού θα πάνε τα χρήματα. Άρα καλό θα ήταν ίσως με τους συντονιστές που θα δώσουν κάποιες κατευθύνσεις να έχουμε ένα έγγραφο εργασίας που θα καθοδηγεί την Επιτροπή μας για τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και ένα δεύτερο έγγραφο εργασίας που θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι αυτές οι αρνητικές προτεραιότητες που κάτι ακούστηκε. Είδαμε να γίνεται κάποιος λόγος, αλλά ε, αυτό που βλέπουμε στο έγγραφο που έχουμε αναχείρες είναι ε, να μας ξεκαθαρίσει η Κομισιόν κάποια πράγματα. Εμείς όμως δεν έχουμε κάποια δουλειά να κάνουμε. Δεν πρέπει να πούμε και εμείς ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Ποια προγράμματα θα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία προσπάθεια να είμαστε ηγετικοί και να δείξουμε σθένος. Δεν θα πρέπει να είμαστε όλο και πιο αδύναμοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ επιθυμώ να εξαγάγω ένα δίδαγμα από τον περσινό χρόνο όπου είχαμε συζητήσει τον προϋπολογισμό του 2011. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε αύξηση 6% και προσπάθησε να την επιτύχει. Στον τύπο και ιδιαίτερα στη Σλοβακία διάβαζε κανείς τότε ότι το διάβημα αυτό των Ευρωβουλευτών ήταν παράλογο. Εγώ θα υποστηρίξω την ε, άποψη του κ. Μπόκρος ότι υπάρχει και το πολιτικό επίπεδο, όχι μόνο το αντικειμενικό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, πάνω από 700 κοινοβουλευτικές εντολές. Βουλευτές δηλαδή. Ο καθένας έχει τη διαφορετική άποψή του. Ο καθένας θέλει να περάσει δικά του πράγματα. Είναι δύσκολο να βρεθούν σημεία όπου μπορούν να γίνουν περικοπές ασφαλώς υπάρχει ένα όριο, περίπου 3% αύξηση των δαπανών. Και το όριο αυτό, το όριο αυτό είναι αυτό μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο προϋπολογισμός του 2012. Βέβαια, στους πολίτες αρέσει να ακούν περί περικοπών στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Την άλλη μεριά όταν γίνονται οι περικοπές δεν τους αρέσει να εφίστανται τις συνέπειες. Και βέβαια οι υπουργοί θέλουν να περικοπούν τα κονδύλια της Ευρώπης, από την άλλη μεριά, δηλαδή αυτά του προϋπολογισμού, από την άλλη μεριά θέλουν να εξασφαλίσουν το δυνατόν περισσότερα χρήματα υπέρ των χώρων τους. Νομίζω λοιπόν ότι το δίδαγμα του 2011 πρέπει να είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε υπερβολικά υψηλές προσδοκίες. Ασφαλώς και είναι σημαντικό να χρηματοδοτηθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι πολίτες των χωρών μας ζητούν να γίνουν περικοπές στο κοινωτικό προϋπολογισμό και το δέχονται. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, πρέπει οι βασικές προτεραιότητες να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ο κύριο ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι γενικά ικανοποιημένο από την έκθεση και θέλω μόνο να μιλήσω για την παράγραφο 66 στην κατηγορία 5. Νομίζω ότι για αυτή τη συνεδρίαση και τον τριμερή διάλογο θα πρέπει να πούμε ότι ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο και να μην λέμε ότι είναι μισοάδιο. Και να σας πω ποιο είναι το νόημα αυτής της έκφρασης. Δεν μπορούμε να πούμε για μια διαπραγμάτευση, για να ξεκινήσουμε μάλλον μια διαπραγμάτευση, πιστεύοντας ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα ε, έχουν κάνει τη δουλειά τους όσον αφορά τις περικοπές, ε, τις διοικητικές δαπάνες, ενώ ε, το Κοινοβούλιο δεν θα έχει κάνει τη δουλειά του. Αντί να πούμε ότι δεν ακολουθήσαμε τη σύσταση του κύριου Επιτρόπου που ζητούσε 1% αύξηση, αυτό αντίθετα πρέπει να πούμε ότι ο προπολογισμό ο δικό μα είναι ένα προπολογισμό λιτότητα. Είναι ένα προπολογισμό που έχουμε κάνει πάνω από 40 εκατομμύρια περικοπέ σε σχέση με την αρχική πρόταση. Ε, έχουμε μία αύξηση, είναι μια τιμαριθμική αναπροσαρμογή στην ουσία σε σχέση με τον προπολογισμό και δεν μπορούμε να πάμε σε μία συνεδρίαση λοιπόν ευάλωτη Ότι δηλαδή δεν τα καταφέραμε να μείνουμε στο 1% και να ακολουθήσουμε το όσα μας ε, είπε ο Επίτροπος. Κάναμε όμως ό,τι μπορούσαμε ώστε να μπορέσει ο προπολογισμό δεδομένων των αρμοδιοτήτων που έχουμε, των υποχρεώσεων που έχουμε και του όγκου του προπολογισμού που έχουμε, ε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επιτύχουμε αυτόν ε, τον στόχο. Κάναμε το, τα μαθήματά μας με τον ίδιο τρόπο που η Κομισιόν και το Συμβούλιο έκαναν και τα δικά τους μαθήματα με βάση τις ισχύουσες συνθήκες. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να παρουσιποβάλουν ένα προπολογισμό που ταυτόχρονα είναι λιτότητας αλλά είναι και Προπολογισμό που να στέκεται στο ύψο ε, το στόχο της ε, νομοθετική ε, αρεστίας, της απαραίτητη πρόβλεψης, ώστε να μπορεί και το Κοινοβούλιο να κάνει τη δουλειά του σωστά. Το κόστος της μη νομοθεσία ή της κακή νομοθεσία είναι και αυτό ένα θέμα που θα πρέπει μία ημέρα των ημερών να μα απασχολήσει και επανειλημμένως θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέσα, όπως σας είπα, ώστε να κάνουμε τη δουλειά που περιμένουν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να ευχαριστήσω λοιπόν την συγγήτρια είναι ακόμα μια μικρή προειδοποίηση ε, για να μην φτάσουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, λες και είμαστε εμείς ε, λάθος έχουμε κάνει όπως σας είπα τα μαθήματά μας και έχουμε φτάσει στο όριο των όσων μπορούσαμε να καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ο Γκέραν Φέρμα ζήτησε και πάλι το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που ξαναπαίρνω το λόγο αλλά άκουσα διάφορα πράγματα για τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσω. Καταρχήν για τον Τζέιμ Άλλη και κάποιου άλλου για τι οικονομικέ εξελίξει. Εγώ πραγματικά και μιλάω πολύ σοβαρά. Δεν νομίζω ότι η μονόχνοτη λιτότητα είναι ο τρόπο να βγούμε από την κρίση. Γιατί η ακραία λιτότητα προκαλεί νέο κόστο βασικά για την μακροπρόθεσμη απασχόληση αλλά και παρεμποδίζει την οικονομική ανάκαμψη. Βλέπω όλα ένα και περισσότερε οικονομίε, κυρίω τα συντηρητικά, συγγνώμη, ε, κυρίως στα συντηρητικά περιοδικά και έντυπα που προειδοποιούν ότι οι ακραίες περικοπές θα κάνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα ιδιαίτερα για την Ελλάδα και την Πορτογαλία που θα, γίνει, θα καταστεί αδύνατο να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους. Δεν είναι ο μόνος τρόπος να βγούμε από την κρίση κόβοντας τα πάντα όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες. Αντίθετα, νομίζω ότι πρέπει να πούμε πως υπάρχουν στρατηγικές προτεραιότητες που είναι σημαντικές για την οικονομική ανάκαμψη σήμερα και ιδιαίτερα οι επενδύσεις για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Και κάποιε από αυτέ τι προτεραιότητε θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και από το δικό μα προπολογισμό. Δεύτερον, αρνητικέ ε, προτεραιότητε. Εγώ είμαι ανοιχτό για κάτι τέτοιο και για μια τέτοια συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που κυρίω υπερασπίζονται τι περικοπέ ε, θα πρέπει να καταστούν υπεύθυνοι για την υποβολή των προτάσεών τους. Οι, οι γραμμικές τώρα περικοπές είναι το αντίθετο των περικοπών των ε, προτεραιοτήτων, συγγνώμη. Όταν προσπαθούμε να πούμε ότι ένα πράγμα είναι πιο σημαντικό από κάποιο άλλο, οι γραμμικέ περικοπέ θα περιέκοπταν και την έρευνα και την ανάπτυξη. Πολύ σημαντικά και στρατηγική σημασία θέματα. Αν το Συμβούλιο λοιπόν είναι έτοιμο να προτείνει περικοπέ στην κοινή γεωργική πολιτική ή περικοπέ στην πολιτική συνοχή σε τομεί που να είναι έτοιμοι να πούνε ναι, συγγνώμη, αυτά τα προγράμματα, δεν δουλεύουν, ε, και είμαι έτοιμο να το συζητήσω. Αλλά κάνουν τι προτάσεις, γιατί αυτοί κυρίω μιλάνε για περικοπές, μάλλον να κάνουν τις προτάσεις αυτοί που μιλάνε για περικοπές και άλλες περικοπές του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόκρο. Θέλει να συνεχίσει το διάλογο. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά ο Γιώργο Φέρμα απευθυνόταν σε μένα. Είμαι ευγνώμων ε, για τις διαλέξεις του για την οικονομία, αλλά δεν είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος και χρόνος για κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να καταστήσω κάτι σαφές. Κανείς δεν υποστηρίζει γραμμικές περικοπές, περικοπές δηλαδή για όλα. Μην με παρεξηγείτε παρακαλώ. Λέω μόνο, λέμε μόνο και ίσως θα μπορούσα να αναφερθώ και σε κάποιους άλλους που είπαν παρόμοια πράγματα. Λέμε μόνο πως το γενικό 4, γενική αύξηση 4,9 ε, δεν θα είναι ρεαλιστική. Καταρχήν, ε, λόγω της αντίστασης της δικής σας ε, κυβέρνησης από τη Σουηδία. Μπορεί να λέτε ότι δεν κατανοώ την πραγματικότητα. Σίγουρα μπορείτε να μιλήσετε πιο μεγαλύτερη εφράδια και να διατυπώσετε καλύτερα τα λόγια σας λέγοντας ότι έχω διαφορετική ερμηνεία. Αλλά φυσικά όλοι μας έχουμε το δικαίωμα να ερμηνεύουμε την πραγματικότητα με διαφορετικούς τρόπους. Δεν πρόκειται για γραμμικές όπως σας είπα περικοπές, αλλά ακριβώς όπως είπε και ο κύριος Έλλης θέλουμε να τονίσουμε τις θετικές και τις αρνητικές προτεραιότητες. Και φυσικά αυτό είναι καταρχήν καθήκον της Επιτροπής ΣΟΥΡ <clears throat> και εκεί ε, πρέπει να τονίσουμε τι, τι πιστεύουμε περισσότερο μακροπρόθεσμα, αλλά πάντως είναι σαφές ότι μια τέτοια γενική υψηλή αύξηση είναι μη ρεαλιστική. και δεν θα το πετύχουμε μέχρι τότε, δεν θα το κρατήσουμε μάλλον μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Καλύτερα είναι από νωρί να είμαστε ρεαλιστικοί και να σχηματίσουμε ρεαλιστικέ και τακτικές προσεγγίσει, ώστε να πετύχουμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κανεί δεν κάνει μαθήματα εδώ οικονομία σε κανέναν άλλο. Παρ' όλα αυτά, εμένα με ενδιαφέρει να διεξαχθεί μια πολιτική συζήτηση ουσίας. Και αυτό γίνεται. Τώρα, λίγα προσωπικά σχόλια, αν μου επιτρέπετε, πριν να δώσω πάλι τον λόγο στην ε, Φρανσέσκα για να συναγάγει τα συμπεράσματα. Συνήθως ακολουθώ τις ε, συμβουλές του James Ellis. Ε, επανέρχομαι τώρα από τις Ηνωμένε Πολιτείες, όπου μπόρεσα να συναντηθώ και με το Κογκρέσο αλλά και με οικονομολόγους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δύο πράγματα βρήκα ενδιαφέροντα. Οι οικονομολόγοι βρίσκονται σε απόλυτο σκοτάδι σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας για τα επόμενα χρόνια σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Είναι, οι γνώμες τους δίστανται. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται λιγότερες δαπάνες, να μειώνονται τα χρέη, να μειώνονται τα ελλείμματα, ταυτόχρονα να υποστηριχθούν οι επενδύσεις για το μέλλον. αυτό τι σημαίνει τώρα σε ό,τι αφορά την επιλογή των δαπάνων, δαπάνες που αυξάνονται, δαπάνες που μειώνονται, τι, τι σημαίνει σε ό,τι αφορά τη σταδιακή προσέγγιση μέσα στον χρόνο για την έξοδο από τη λιτότητα. Εκεί οι γνώμες τους δίσταται και ουδής γνωρίζει ακριβώς. Καμία χώρα, ή μάλλον ορισμένες χώρες έχουν βρεθεί στην κατάσταση αυτή εδώ και ορισμένα χρόνια, αλλά ποτέ δεν υπήρξε αυτή η συγκυρία, συγκυρία ε, περιστάσεων σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Άρα δεν υπηρξε αυτη η συγκυρια συγκυρια περιστασεων σε ολο Το ανεπτυγμενο κοσμο αρα δεν ξερουν Το δεύτερο που με εξέπληξε είναι ότι πολιτικά η νοοτροπία συνεχίζει να λέει μείωση των ελλημάτων, μείωση των δαπανών κτλ. Ταυτόχρονα η συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες που μπαίνει σε, σιγά σιγά σε προπαρασκευή της προεκλογικής εκστρατείας για του χρόνου λέει ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα είναι της τάξης των 4-3 εκατομμυρίων δολαρίων εξοικονομήσεις δηλαδή που προτείνει ο πρόεδρος Ομπάμα ή 6-3 ε, εκατομμύρια δολάρια που προτείνει ο ομόλογός μου, πρόεδρος δηλαδή, Πολ Ράιαν, πρόεδρος της ε, ε, Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκεί βέβαια αυτός έχει και περισσότερη εξουσία από τον ίδιο τον πρόεδρο των Ενωμένων Πολιτειών που όπως γνωρίζετε το σχέδιο προϋπολογισμού επί του οποίου γίνεται συζήτηση και εγκρίνεται δεν είναι αυτό που υποβάλει ο πρόεδρος της, ε, των ΗΠΑ, αλλά τα κοινοβουλευτικά σώματα. Να λοιπόν αυτή είναι η ε, σκέψη τους ακόμα και, και σε πολλές χώρες μέλη επίσης δικές μας. Οι συνάδελφοι που υπενθυμίζουν το πολιτικό αυτό πλαίσιο έχουν δίκιο που το υπενθυμίζουν τη στιγμή που αρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών πρέπει να μην ότι όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί σε όλες τις χώρες μας έχουν ένα είδος έμμονης ιδέας να μειώσουν δηλαδή τις δαπάνες. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την άποψή τους, αλλά πάντως πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η σκέψη τους. Θα ήθελα εγώ τώρα να επαναλάβω τρεις ε, συστάσεις ε, τακτικού χαρακτήρα. Πρώτη, θα πρέπει να αγωνιστούμε πολιτικά, πολιτικά στην, στην ε, πολιτική διαπραγμάτευση για τις ε, ε, πιστώσεις υποχρεώσεων και όχι πληρωμών. Το λέω αυτό, το επαναλαμβάνω, το έχουμε ξεχάσει. Το ξαναλέω. Πολιτικά αυτό που είναι σημαντικό είναι οι πιστώσεις υποχρεώσεων. Από τη στιγμή που αναλαμβάνει κανεί μια υποχρέωση είναι και υποχρεωμένο να πληρώσει. Πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε και στο Συμβούλιο και στον τύπο και στην κοινή γνώμη ότι όταν, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση των πιστώσεων πληρωμών είναι επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Βέβαια, για τα Υπουργεία Οικονομικών των χωρών μελών για αυτά που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτά μετρούν. Από την άποψη πολιτική όμως, επαναλαμβάνω ότι είναι οι πιστώσεις υποχρώσεων εκείνες. Διότι οι πιστώσεις πληρωμών και απολογιστική άποψη λαμβάνεται η απόφαση τη στιγμή που λαμβάνονται αποφάσεις για τις πιστώσεις υποχρώσεων. Αυτό μου φαίνεται λοιπόν ότι είναι σημαντικό και που πρέπει να υπομνηστεί. Δεύτερη σύσταση. πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλέσουμε τους Υπουργούς Οικονομικών και ιδεοδός, ελπίζω, και τους εθνικούς ηγέτες να συγκρίνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς με τον ευρωπαϊκό. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζω απολύτως την εξαρχής προσέγγιση της Φρανσέσκα να προσπαθήσει δηλαδή να συνδέσει την διαδικασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με τη νέα διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου που ενισχύει την, τον συνδυασμό των ε, εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. Γιατί και στους εθνικούς προϋπολογισμούς γίνεται προσπάθεια μείωσης των δαπανών. Ωστόσο παρόλα αυτά ορισμένες δαπάνες αυξάνονται. Φυσικό είναι αυτό. Και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει μια σύνθεση απόλυτα διαφορετική από αυτή των εθνικών προπολογισμών, όπου οι μισές δαπάνες είναι λειτουργικές, είναι δηλαδή μισθή των υπαλλήλων, ενώ εδώ είναι μονάχα 6%. Το μέγα μέρος του προϋπολογισμού μας διατίθεται είτε σε οικονομικές παρεμβάσεις είτε σε επενδύσεις. Πρόκειται λοιπόν για κεφάλαια που και στους εθνικούς προϋπολογισμούς μειώνονται λίγο ή λιγότερο εν πάση ή καμιά φορά τα αυξάνουν κιόλα. Αν θέλουμε λοιπόν τώρα να πείσουμε του ε, ε, υπουργού οικονομικών ότι πρέπει να εξετάσουν τον κοινοτικό προπολογισμό με διαφορετικό μάτι από αυτό με, τον, με το οποίο εξετάζουν τους εθνικούς του προπολογισμού, θα πρέπει να τους ζητήσουμε να ε, προχωρήσουν με τον τρόπο αυτό. Τρίτη σύσταση, πάλι δεν είναι νέα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπομνηστεί, είναι να δείξουμε επίσης στους υπουργούς, στους υπουργούς οικονομικών των χωρών μελών, ότι δεν είναι επειδή ορισμένες χώρες μέλη και όχι όλες ε, έκαναν μια πάρα πολύ άσχημη διαχείριση, δηλαδή πέταξαν τα λεφτά τους από το παράθυρο. Δεν σημαίνει ότι τώρα για το λόγο αυτό πρέπει να γίνουν δραματικές εξοικονομήσεις, ότι δηλαδή πρέπει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει για κάποιες χώρες που έκαναν άσχημη διαχείριση. Αν ορισμένες χώρες οφείλουν να προχωρήσουν σε σημαντικότατες εξοικονομήσεις, αυτό οφείλεται στην κακή διαχείριση, διότι ακριβώς κατασπατάλησαν τα χρήματά τους τα προηγούμενα χρόνια. Αυτές οι χώρες λοιπόν δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, άρα πρέπει αυτός να πληρώσει. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, επιστρέφοντας σε έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό που θα χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Διότι όσο δεν χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους θα είμαστε βέβαια όμοιροι των χωρών που έκαναν την χείριστη διαχείριση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επιθυμίζουμε διαρκώ, διότι η εμπειρία δείχνει ότι όταν, το λέμε αυτό μια πρώτη φορά στον τριμερή διάλογο, κανένα δεν μα ακούει. Όταν το λέμε σε ένα τέρι φορά, μα ακούν αλλά δεν αντιδρούν και όταν το λέμε τρίτη φορά, μας ακούν, αντιδρούν αρνητικά. Και ε, μετά προχωρήστε. Τέσσερις-πέντε φορές, ίσως κάποια στιγμή να δούμε και μια αντίδραση θετική. Τελευταίο τώρα σχόλιο σχετικά με την τακτική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Το προηγούμενο έτος, απέναντι στο Συμβούλιο, δοκιμάσαμε μια ασυνήθιστη τακτική σε σχέση με τα όσα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις περί προϋπολογισμού. Εγώ ο ίδιος μάλιστα είχα ταχθεί υπέρ αυτής της ασυνήθιστης τακτικής. Η τακτική αυτή έγκυτο στο να πούμε αρκετά νωρί, όχι στην πρώτη ψηφοφορία, αλλά πάντως αρκετά νωρί, ότι ήμασταν διατεθειμένοι να έλθουμε στην, στην θέση του Συμβουλίου, στο ποσό του Συμβουλίου δηλαδή, χωρίς να προσθέσουμε τον ευρώ. Και εκεί το Συμβούλιο έκανε κάποιες πολιτικές παραχωρήσεις. Αυτή η τακτική δεν επέτυχε. Θα δούμε τώρα ποια τακτική θα μας προτείνει η συγκεντριά μας. Αλλά εν προκειμένου, σε αυτή δηλαδή την περίοδο του έτους, σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων θα έλεγα να επανέλθουμε στην προηγούμενη τακτική που είναι τακτική αντιπαράθεσης αντιπαράθεσης επί του ετησίου προπολογισμού όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβάλλει αριθμούς, νούμερα, αριθμητικά στοιχεία διαφορετικά από αυτά του Συμβουλίου. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχουμε συνείδηση του γεγονότος ότι εάν θέλουμε να, είμαστε, να έχουμε θετικό για μας συσχετισμό δυνάμεων με το Συμβούλιο όπως έχουν πει και πολλοί από εσά, θα πρέπει να είμαστε ικανοί να προτείνουμε και αρνητικές προτεραιότητες. Εάν τοποθετηθούμε σε μια διαπραγματευτική θέση όπου θα πούμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε όλες, όλα τα κονδύλια, όλες τις γραμμές του προϋπολισμού, θα, η θέση μας δεν θα είναι πολύ ισχυρή πολιτικά, εάν ωστόσο δείξουμε ότι Έχουμε κατανόηση για την θέση του Συμβουλίου, ότι είμαστε διατεθειμένοι να την λάβουμε υπόψη και ότι ταυτόχρονα επιθυμούμε κάτι που μας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο για το μέλλον δηλαδή και υπόψη, έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και τι νέε αρμοδιότητε που δίνει η Συνθήκη τη Λισαβόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θέλουμε να αυξήσουμε ορισμένα κονδύλια, ενώ από την άλλη μεριά είμαστε διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουμε τι αυξήσεις αυτέ τουλάχιστον εν μέρη, με μειώσει, με εξοικονομήσει αλλού. Εάν θέλουμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να, κάνουμε, να είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εξοικονομήσεις σε κονδύλια τα οποία θα θίξουν το Συμβούλιο. Και τότε θα μας ακούσουν βέβαια. Διότι και κάθε χρόνο γίνονται εθνικές εκλογές σε 6-7 χώρες μέλη στατιστικά. Του χρόνου για παράδειγμα ε, υπάρχουν εθνικές εκλογές στη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία αλλά και άλλες. Εάν κάποια στιγμή το φθινόπορο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδείξει ότι σε ορισμένα κονδύλια προχωρεί σε περικοπές της τάξης του 5, 10, 20% σε κονδύλια που ενδιαφέρουν τις χώρες αυτές πολύ, τότε θα είναι διαφορετική η κατάσταση, θα είναι διαφορετική και η θέση μας. Αυτή λοιπόν είναι, αυτές είναι μάλλον οι παρατηρήσεις, οι συστάσεις που κάνω. Βεβαίω, τώρα το λόγο θα λάβει η Φραντσέσκα για να συνοψίσει. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και θα πω στους συναδέλφους ότι αυτό το κείμενο οπωσδήποτε έπρεπε να εμπλουτιστεί με τη συμβολή τους και κυρίως θα πρέπει να συμπληρωθεί με τα συμπεράσματα που θα ήθελα όντω να προέλθουν από τη συζήτηση και από τις προτάσει τροπολογίες που θα καταθέσουν οι συνάδελφοι και οι πολιτικέ ομάδες. Ωστόσο θα ήθελα κάτι πολύ βασικό να ξεκαθαρίσω. Μέσα σε αυτό το κείμενο ποτέ δεν εξέφρασα τη λύπη μου για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις. Απλώς έχω προσπαθήσει να εντοπίσω όσο γίνεται με μεγαλύτερη διαφάνεια αυτά που δεν είναι αυξήσεις. Αναφέρομαι για παράδειγμα στις αυξήσεις των ταμείων που σχετίζονται με την πολιτική μετανάστευση. Δεν πρόκειται για πολιτικές ή θελημένες στρατηγικές αυξήσεις μέσα στην πρόταση της Κομισιόν για τον προπολογισμό 2012 σε απάντηση στις επίγουσες ανάγκες. Συνδέω συνδέονται με τον προγραμματισμό 2007-2003. Άρα πρόκειται για ενημέρωση και για να αναπροσαρμογή απλώς. Νομίζω λοιπόν ότι το σημείο κίνησης για κάθε συζήτηση και για την επεξεργασία εν γνώση των, ε, θεμάτων ε, της θέσης μας θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποιο είναι το status quo. Να αποσυνθέσουμε αυτά δηλαδή που να είναι αυξήσεις και να τα τοποθετήσουμε μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικών προπτικών 2007-2013 για να δούμε αν είναι όντως πολιτικές αποφάσεις ή αν είναι αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από 5 χρόνια. Και ε, εδώ σε κάποιο παράγραφο λέω ότι ένα πακέτο του προγράμματος ΣΥΠ, ε, ε, ΤΕΝ, ενεργειακά δίκτυα κτλ. Αυτά δεν αφορούν την στρατηγική 2020. Αποτελούν καρδιά μεν της στρατηγικής 2020 αλλά θα υποχρηματοδοτηθούν σε σχέση με τα όσα είχαν αποφασιστεί το 2006 και για το πακέτο 2007-2013. Είναι στην ουσία ή θα έχουν πάρει μια πολύ μικρή ε, αύξηση ίσα ίσα δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε σε επικρίσεις και προτάσεις βελτίωσης, θα πρέπει να έχουμε τις σωστές πληροφορίες στη διάθεσή μας. Και αυτό σημαίνει, όσον αφορά τα νούμερα, ε, πληροφορίες που να έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Μπορεί κανείς να πει το, να μία κατάφαση και την αντίφαση της στην ίδια στιγμή για όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με, το πέρσι, με την περσινή χρονιά είναι αλλαγές που είτε εντάσσονται στο πολιετές πλαίσιο είτε πρόκειται απλώς για προσαρμογή του πολιετούς προγράμματος. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω, όπως νομίζω πως κατά κάποιο τρόπο ξεκαθάρισα στη συζήτηση που ήδη κάναμε για τις προτεραιότητες ότι η δική μου προσωπική θέση είναι αντίθετη όχι μόνο στις οριζόντιες περικοπές αλλά και στις οριζόντιες αυξήσεις. Αυτό που δεν θέλουμε και που δεν είναι σκόπιμο δεν είναι μόνο μια μαθηματική μείωση αλλά και μια μαθηματική αύξηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Είναι το λιγότερο ευρωπαϊκό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Αυτό που είναι απαραίτητο αντίθετα να τονίσουμε είναι ε, μια στρατηγική επιλογή. Δηλαδή η βούληση να χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό για να τον καταστήσουμε ένα ζωντανό μέσο που ε, επηρεάζεται και αντιδρά στους καιρούς και στις καταστάσεις. Και γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε με τη στρατηγική 2020. Γιατί αν η στρατηγική 2020 ήδη είχε χρηματοδοτηθεί από το 2006 και είχε προβλεφθεί, τότε διερωτώ τι συζητήσαμε πέρσι όταν την ορίσαμε και την καθορίσαμε και την αποφασίσαμε στο Κοινοβούλιο. Δεν, είναι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο λοιπόν. Δεν μπορεί να έχει προβλεφθεί από το 2006. Ελπίζω πως όχι δηλαδή. Άμα θέλουμε αυτή η στρατηγική του 2020 να αποτελέσει μια, ένα μέσο για διέξοδο από την κρίση, θα πρέπει να ε, την χρηματοδοτήσουμε αυτή τη στρατηγική για να μπορέσει να ενοφέλουμε με προσεκτική χρήση του προϋπολογισμού, με αυξήσεις, περικοπές, όχι μαθηματικού τύπου, αλλά στρατηγικού τύπου με βάση μια σαφή ανάγνωση των ε, επιλογών για το 2012 σε σχέση με τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές και επίσης ξεκινώντας από ένα βασικό στοιχείο ότι δηλαδή ναι έχουμε ένα προπολογισμό που αποτελείται από υποχρεώσεις και πληρωμές αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όσον αφορά τις πληρωμές ε, όπως έλεγα και στην εισήγησή μου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά τις προβλέψεις των κρατών μελών γιατί τα κράτη-μέλη είναι αυτά που στο Συμβούλιο Συμβούλιο κρατούν διαφορετικές θέσεις, αλλά που διαχειρίζονται και το 80% του προπολογισμού μας. Συμμερίζομαι απόλυτα την ιδέα του να έχω, δώσουμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτές τις αρνητικές προτεραιότητες, δηλαδή να αρχίσουμε να εστιάζουμε στο ποιες θα μπορούσαν να είναι οι αρνητικές προτεραιότητες που θα πρέπει να τις αναγνώσουμε με υπό το φως των θετικών προτεραιοτήτων του Συμβουλίου και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω πως το ίτερ στην πρόταση ψηφίσματός μου η θελημένα έχει ενταχθεί εδώ ως ένα σημείο πολύ λεπτό στις ε, ε, διαπραγματεύσεις. Δηλαδή είναι κάτι το πολύ ανοιχτό και εδώ θέλω να απαντήσω έτσι στον συνάδελφο ε, Άγκλουντ και στον συνάδελφο Τρούπελ. Είναι πολύ ανοιχτό αυτό το θέμα στην πρότασή μου και μπορούμε να και ανοιχτό σε διαπραγμάτευση. Ε, εντό εισαγωγικών. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από μια διαφανή ανάγνωση της ε, πρόταση Κομισιόν που βασίζεται στις δημοσιονομικέ προπτικές και ήθελα με την ομάδα εργασίας να καθορίσουμε τις δικές μας στατικές προτεραιότητες πολύ σοβαρά σε σχέση με τις προτεραιότητες 2020 και να προσπαθούμε να δούμε τι θέλουμε, τι θέλουμε ως καινοτομία σε αυτό το προπολογισμό σε σχέση με τις επιλογές που κάναμε πέρσι και τι οποίε ε, πρέπει πλέον να αρχίσουμε να θέτουμε, θέτουμε σε εφαρμογή. Γιατί αν θέλουμε, αν όντω μάλλον ε, αυτή η στρατηγική του 2020 να αρχίσει να χρηματοδοτείται με την αρχή των νέων δημοσιονομικών προοπτικών, θα έλεγα ότι χάσαμε το μισό χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μα για να θέσουμε σε εφαρμογή. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και εγώ την Φραντσέσκο όσον αφορά αυτή την εντολή διαπραγμάτευση για τον τριμερή διάλογο. Έχουμε προβλέψει μια ακόμα ανταλλαγή απόψεων επί τη βάση του συμπληρωματικού κειμένου που μας ε, είπε η Φραντσέσκο ότι θα μας δώσει για την ε, συνεδρίαση της 23 και 24 Μαΐου. Η ημερομηνία για, η διορία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 24 Μαΐου το μεσημέρι και η έκθεση θα πρέπει να υιοθετηθεί στην Επιτροπή Προπολογισμού στις 15 Ιουνίου με στόχο να υιοθετηθεί στην Ολομέλεια τον Ιούλιο ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον τριμερή διάλογο του Ιουλίου. Ε, να προτείνω τώρα να περάσουμε στο σημείο 8 της ημερήσιάς μας διάταξης. Συνάδελφος Άγκλουντ θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του για το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρατόμ. Συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας εκθέσω τις αρχικές μου ιδέες σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο Ευρατών. Πρόκειται για ένα θέμα που καθήλυνα αρμόδια είναι η Επιτροπή Ήτρε, αλλά δεν είναι ακόμα πλήρως καθορισμένο και το χρονοδιάγραμμα. Ίσως θα μπορούσαμε αυτό το θέμα το συζητήσουμε τα μέσα Ιουνίου, οπότε και θα έχω μάλλον έτοιμο το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Όπως είπα στην προηγούμενη παρέμβασή μου, το βασικό θέμα είναι το ίτερ και πώς θα λύσουμε τα χρηματοοικονομικά προβλήματα. Αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον θέμα. Ουσιαστικά συζητούμε για ένα πρόγραμμα πλαίσιο το 2012-2013 γιατί δεν, επιλέ... δεν ε, υπάρχει δυνατότητα για προγράμματα πάνω από πέντε χρόνια. Ουσιαστικά μιλάμε για επέκταση των προγραμμάτων που ξεκίνησαν το 2007 και θα λήξουν φέτος. Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για το οποίο συζητούμε λοιπόν. Έχω αναλάβει λοιπόν τη σύνταξη της γνωμοδότησης. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για μας να υπογραμμίσουμε για μια ακόμη φορά το γεγονός ότι θεωρούμε και ελπίζω να συμφωνήσουν περισσότεροι μαζί μου. Θεωρούμε λοιπόν ότι η τρέχουσα ρύθμιση ότι δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στην διοίκηση ΙΤΕΡ της ε, Ευρατόμ που καλούνται να λάβουν τις ε, αλλά εμείς καλούμαστε να, να λάβουμε τις δύσκολες αποφάσεις για την ε, χρηματοδότηση αυτής της δραστηριότητας. Νομίζουμε ότι δεν είναι σωστή αυτή η ρύθμιση, αυτή η διευθέτηση. Άρα Νομίζω ότι στη γνωμοδότηση αυτή μπορούμε να το ζητήσουμε. Θέλουμε μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο και υποπτία της δραστηριότητας αυτής για να διευκολύνουμε και τις μελλοντικέ δύσκολε αποφάσει που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα. Αναπόφευκτα προκύπτει και το ζήτημα του πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτός ο αντιδραστήρας, ε, το ίτερ δηλαδή, αυτή είναι η βασική δραστηριότητα του προγράμματος. Εδώ έχουμε την πρόταση της Κομισιόν. 100 εκατομμύρια το 2012 και 360 εκατομμύρια για το 2013. Τα λέει και η έκθεση της Φραντσέσκα για τον προπολογισμό του επόμενου έτους, αλλά έχει να κάνει και με την έκθεση του Ράιμερ Μπέγκε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα και οι τρεις μας καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση. Δεν είμαι ικανοποιημένο με τον τρόπο που προτείνει η Κομισιόν για επίλυση αυτού του ζητήματο. Και νομίζω ότι και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, αλλά και σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε που είπα καθήλυνα αρμόδια είναι η Επιτροπή Ήτρε, εγώ δεν έχω να πω πολλά πάνω σε αυτό. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Έχουμε όμως τα δημοσιονομικά ζητήματα. Που μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως προείπα, από πέρυσι είδαμε ότι υπήρξαν μη εκμεταλλευτήσεις πιστώσεις Κατά την άποψή μου ήταν πολύ δημιουργικό το Συμβούλιο και βρήκε μια λύση για το πώς μπορεί να, να χρηματοδοτηθεί το ΙΤΡΕ. Αν υπήρχε πολιτική βούληση, θα μπορούσε η ρύθμιση να γίνει πολύ διαφορετικά σε ό,τι αφορά τις μη εκμεταλλευτήσεις ε, πιστώσεις. Θα μπορούσαν ε, βέβαια να δοθούν τεχνικές εξηγήσει για το πώς αυτό δεν είναι εφικτό κτλ. Αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι αν υπάρχει ε, θέληση υπάρχει και τρόπος. Είμαι πεπισμένος ότι δεν υπάρχει θέληση. Άρα η προτινόμενη λύση και πάλι θα ροκανίσει το 7ο πρόγραμμα. Και υπό το πρίσμα και της Αντιγικής 2020 είναι πολύ κακή η λύση κατά την άποψή μου. Πολύ κακή είναι η λύση και καθαρά από πλευράς του πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα προπολογισμό και του πώς ε, επίσης μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις εξουσίες που έχουμε. Κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να δούμε στην γνωμοδότηση αυτή είναι ότι ίσως θα έπρεπε κάπως να περιχαρακώσουμε αυτή την ε, ε, χρηματοδότηση δραστηριότητα για το μέλλον. Δηλαδή να έχουμε βάλει κάποια όρια να μην βρεθούμε στην ίδια κατάσταση. Να προκύψει μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική αντιπαράθεση όσο σημαντικότερη. Ήδη ξέρουμε τι γίνεται εδώ και ένα χρόνο περίπου και δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα. Άρα είναι και αυτό ένα θέμα σημαντικό. Κάτι άλλο που σχετίζεται ακριβώς με το ότι δεν έχουμε τον έλεγχο που θα θέλαμε να έχουμε στο πλαίσιο της όλης αυτής της διαδικασίας εφόσον εμείς είμαστε που πρέπει να εξεύρουμε τη χρηματοδότηση για αυτή τη δραστηριότητα, φαίνεται ότι η Κομισιόν να μην θέλει να προβεί σε μια πραγματική εκτίμηση επιπτώσεων του προγράμμα, των προγραμμάτων που θα, του προγράμματος μάλλον που θα λήξει φέτος, πεντέτους προγράμματος. Από τεχνικής πλευράς απλά θα παραταθούν για δύο ακόμα χρόνια, 2012 και 2013, τα προγράμματα. Αυτό ναι, αληθεύει από τη μία, αλλά από την άλλη πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο προπολογισμό για όλο αυτό το έργο και την όλη δραστηριότητα δεν ήταν επαρκής. Ή τέλο πάντων ε, δεν ήταν ε, πλήρης αξιοποίηση των κονδύλων. Άρα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση επιπτώσεων. Τώρα η Επιτροπή ε, θα πάει στη Γαλλία, μια αντιπροσωπεία της έχουμε λάβει κάποια έγγραφα στη διάθεσή μας. Δεν ε, θα είμαι εγώ στην αντιπροσωπεία, αλλά θα μελετήσω αυτά τα έγγραφα. Ελπίζω πάντως όσοι πάνε στην αντιπροσωπεία στη Γαλλία, με την αντιπροσωπεία στη Γαλλία να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες που θα πρέπει να τους λάβουν υπόψη μας και στην τελική γνωμοδότηση που θα εκπονήσω εγώ. Τέλος, και επανέρχομαι κύριε Πρόεδρε, στα όσα έγιναν στην Ιαπωνία πολύ πρόσφατα. Η πυρηνική ασφάλεια είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να επισημάνουμε. Άλλωστε εντάσσεται η πτυχή αυτή στο πρόγραμμα πλαίσιο Ευρατόμ και νομίζω ότι είναι κάτι που απασχολεί τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν επαρκείς οικονομικοί πόροι για να μπορέσουμε να εστιάσουμε στην πυρηνική ασφάλεια. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε στο πλαίσιο της γνωμοδότησης. Αλλά στα πιο λεπτομεριακά θα αφήσουμε να γνωμοδοτήσει η Καθήνα Αρμούδια Επιτροπή Ήτρε. Σας εξέθεσα τι ε, σκοπεύω να συμπεριλάβω στη γνωμοδότησή μου και προσβλέπω στα σχόλιά σας αλλά και όπως είπα πριν στην καλή συνεργασία με τη Φραντσέσκα και τον Ράιμερ για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση και να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την επίλυση του ζητήματος και μια καλύτερη, ένα καλύτερο προσανατολισμό της διαδικασίας σε σχέση με αυτήν που έχουμε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα. Όπως είπατε, έχουμε την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών που θα πάει στο Κανταράς της Γαλλίας σε ένα εργοτάξιο ουσιαστικά, ε, εκεί που θα έχουμε το ερευνητικό κέντρο ΙΤΕΡ. Και πιστεύω ότι θα έχουμε ενημέρωση από τους συναδέλφους που θα μεταβούν στο Κανταράς όταν επιστρέψουν. Και βέβαια σίγουρα μετά την καταστροφή στην Ιαπωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε όλους τους πυρηνικούς σταθμούς ε, που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους υποβάλει σε τεχνικές δοκιμές αντοχής ε, αν μπορούν να θέξουν οποιοδήποτε είδους ατύχημα που σχετίζεται με το κλίμα, με τη γεωλογία, με ανθρώπινο σφάλμα κτλ. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στο βαθμό που βέβαια αυτά τα stress test, αυτές οι δοκιμές αντοχής ε, θα έχουν αποτελέσματα τα οποία θα μπορούμε να τα έχουμε πριν την εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτος ο κύριος Ντέρεκ Βόν. Ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Χάγκλουντ για την εισαγωγή που έκανε στο σχέδιο γνωμοδότησής του. Δεν είμαι αντίθετος με τα πυρηνικά θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου έτσι κι αλλιώς με τον τρόπο αυτό. Όπως είπε βέβαια ο κύριος Χάκλουντ, πρέπει να διασφαλίσουμε και την ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως εκ τούτου πρέπει να διδαχθούμε και τα μαθήματα από την πρόσφατη καταστροφή στην Ιαπωνία για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης όμως και για την εκπαίδευση του προσωπικού, για την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα πυρηνικής ασφάλειας και ούτω καθεξής. Έρχομαι στο πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω. Την άρση δηλαδή της υποχρέωσης ε, μελέτης επιπτώσεων για το προηγούμενο πρόγραμμα. Όπως είπα πρέπει να διδαχθούμε από τα όσα συνέβησαν και για τον προϋπολογισμό βέβαια και είναι σημαντικό να το εξετάσουμε τουλάχιστον να γίνει μελέτη επιπτώσεων. Αυτό θα ήθελα να συζητηθεί στο προσεχές μέλλον. Επίσης έρχομαι στον ίδιο τον προϋπολογισμό τώρα, μιας και είμαστε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών που αυτό μας απασχολεί περισσότερο στη γνωμοδότηση αυτή, ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι μέσα στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο και οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν το 2011. Έγιναν και συζητήσεις πέρσι, οι συζητήσεις πέρσι στο, ε, για το ΊΤΕΡ και θα συνεχιστούν και στις διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν με τις προτάσεις και όλες που κάνει η Φραντσέσκα στην εκθεσή της. Βλέπουμε επίσης και τις πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την λήψη κονδυλίων από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα για το ίτερ από το, το, στο ύψος των 100 εκατομμυρίων. Εάν το κάνουμε αυτό, θεωρώ ότι θα υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουμε προβλήματα για τη χρηματοδότηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου και επομένως και για την επίτευξη των στόχων του 2020. Αυτά πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη. Εγώ θέλω να ενταχθεί αυτό το θέμα στα, στη διαπραγματεύση για τον προπολογισμό του 2012 και αναμένω βεβαίω και την περαιτέρω πορεία τη γνωμοδότηση του κ. Χάγκλουτ. Η κυρία Γένσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, υποστηρίζω τη γνωμοδότηση του Καρλ Χάγκλουντ. Λαμβάνω το λόγο μόνο για να, να αναφερθώ στην αντιπροσωπεία που θα πάει στο Κανταράς μαζί με τον Μπαρτ Στάις Είμαι επικεφαλής αντιπροσωπείας αυτής, ο Μπατ από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Η πρώτη συνάντησή μας έγινε χθε με εμπειρογνώμονες που εξήγησαν τα τεχνικά θέματα καθώς και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξήγησαν τις οικονομικές πτυχές. Προφορώ την Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι εδώ έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε με σοβαρό και αυστηρό τρόπο. Κάναμε ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και για θέματα ασφαλείας, ε, για θέματα που ίσως προκαλέσουν περαιτέρω κόστος. Η πρώτη εντύπωσή μου από τη χθεσινή συνάντηση είναι ότι όντως θα χρειαστεί να βρούμε τρόπο να διαφυλάξουμε τη χρηματοδότηση. Να φροντίσουμε δηλαδή να τηρηθεί σε πλαίσια η χρηματοδότηση του έργου, διότι δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον. Και εάν δεν θέλουμε να αρχίσει να επεκτείνεται σε άλλους τομείς, όπως βλέπουμε τώρα με το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα υπαριθμών 7, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, όπως είπα, να περιορίσουμε, να, να, ορίσουμε, δηλαδή να μην επιτρέψουμε να ξεφύγουν από κάποια όρια, ε, να ξεφύγει από κάποια όρια το κόστος του ίτερ. Αφού ε, τα χρήματα για το ίτερ πάνε να τα πάρουν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όσο περισσότερα ακούω, τόσο πιο ενδιαφέρον μου φαίνεται το θέμα. Επίσης θέλω να καταστήσω σαφές ότι αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι να δουλέψουμε, όπως είπα, πολύ σοβαρά για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρίπελ. Yes, you will not be as Δεν θα εκπλαγείτε ότι όπου θα σας πω ότι εμείς οι πράσινοι είμαστε αντίθετοι με την πρόταση αυτή για διαφόρους λόγους. Πρώτον, το πρόγραμμα είναι σαφής έκφραση της ε, φιλοπυρηνικής πολιτικής και προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερο, η σημαντική αύξηση των δαπανών για αυτό τον λευκό ελέφαντα που λέγεται ίτερ θα οδηγήσει σε μείωση δαπανών για άλλες ανανεώσιμες ενέργειες. Και μάλιστα σε περίοδο λιτότητας βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην διστάζει να προσθέτει 1,3 δις ευρώ μόνο για το 2012 και 2013 για το έργο αυτό. Για μας αυτό σημαίνει μια ε, απίστευτη έλλειψη ισορροπίας, διότι έχουμε, κάνουμε προσπάθεια για ε, βιωσιμότητα, για ανανεώσιμες ενέργειες. Πάμε τώρα και παίρνουμε 460 εκατομμύρια από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για να τα δώσουμε στο ίτερ. Βρίσκω ότι είναι μια πολύ άσχημη απόφαση αυτή. Δεν οδηγεί στην απαραίτητη αναπροσαρμογή των ενεργειών. Από την άλλη μεριά μπορούμε να δεχθούμε βέβαια χρήματα τα οποία διατίθενται για την πυρηνική ασφάλεια που φαίνεται να είναι πιο σημαντική από ποτέ. Άκουσα πριν τον Τέρεκ για παράδειγμα να λέει ότι πρέπει να συνταχθεί μελέτη επιπτώσεων. Νομίζω και εσείς κύριε Πρόεδρε το είπατε. Χθε όμως άκουσα ότι ο αρμόδιος επίτροπος καθώς και οι άλλοι επίτροποι υπαναχωρούν σε σχέση, ο κύριος Έτιγκερ δηλαδή, υπαναχωρούν ε, σε σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μετακίνηση των ενεργειών. Τώρα έχω ε, και μία ερώτηση σχετικά με τον ορισμό ή περιορισμό των δαπανών. Καλύτερα έτσι βέβαια παρά να ανοίξουμε τις πύλες στη χρηματοδότηση αυτή. Τι θα σημαίνει όμως αυτό το ring fencing τελικά. Θα υπάρξουν ξεκάθαρες γραμμές για την έγκριση του προϋπολογισμού του ίτερ ή υπάρχει κίνδυνος η πλειοψηφία να γιστάσουμε τελικά το έργο αυτό να είναι όπως λέμε ε, στα γερμανικά investitions ruin, δηλαδή ένα επενδυτικό ερήπιο. Να μείνει εκεί δηλαδή μισοφτιαγμένο. Αυτά θα πρέπει να δούμε βέβαια και στο Καταράς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Καβαλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή του που μας έδωσε κάποιες πρώτες ιδέες και να τονίσω τη σημασία του ΙΤΕΡ και επί της ουσίας πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική πηγή ενέργειας που θα είναι καθαρή και προσιτή οικονομικά. Προς το παρόν, καμία από τις πηγές ενέργειας που έχουμε δεν έχει, δεν στερείται μειονεκτημάτων. Άρα είναι πολύ σημαντική η έρευνα αυτή για να βρούμε μια καθαρή και προσιτή οικονομικά πηγή ενέργειας που δεν θα έχει τα μειονεκτήματα της κανονικής διαδικασίας ε, πυρηνικής σύνδεξης, σχάσης. Η θέση μας ε, απέναντι στους εταίρους μας επίσης είναι κάτι που πρέπει να το δούμε στον τομέα της ενέργειας. Για το ΙΤΕ τώρα, ακόμα κάτι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έγιναν κάποια σφάλματα, ό,τι αφορά τη διαχείριση ή την, ε, τις υπερβολικές δαπάνες λόγω του κακού σχεδιασμού της διαχείρισης ακριβώς. Αυτό πρέπει να αλλάξει. και να υπάρξουν ε, νέοι τρόποι, ένα νέο μοντέλο διακυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, Συμφωνώ με συναδέλφους ε, που μίλησαν πριν και είπαν ότι θα πρέπει αυτό το έργο να θέσει σε κίνδυνο άλλες προτεραιότητες ε, του 7ου προγράμματος πλαισίου γιατί έχουμε θέσει μια σειρά προτεραιοτήτων για αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την υγεία, για ενέργειες όπως ε, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ICT, ε, σημαντικές προτεραιότητες για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε με έναν εύλογο τρόπο και με σωστή διοίκηση και διαχείριση να συνεχίσουμε το έργο ITER χωρίς όμως να διακινδυνεύσουμε τους βασικούς στόχους μας, τις βασικές μας προτεραιότητες στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλήσεων. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά πρέπει να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ, Ράιμερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Καρλ Αγγλούτο για το σχέδιο γνωμοδότησης που μας παρουσίασε. Θέλω να τον συγχαρώ και πράγματι είναι καλό να έχουμε μια κοινή προσέγγιση οι τρεις εισηγητές. Σκεπτόμενος αυτά που είπαμε και χθες στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση της αντιπροσωπείας που θα μεταβεί στο Κανταράς, πρέπει να αναγνωρίσω ότι ότι οι γενικοί διευθυντές της Κομισιόν και οι τρεις εκπρόσωποι των ε, ερευνητικών ε, ε, κύκλων ε, μετά από όσα μας είπαν, πρέπει να δούμε το εξής. Θα μας πει βέβαια η αντιπροσωπεία μετά. Το θέμα είναι πώς θα δράσουμε πολιτικά απέναντι σε αυτά τα πολύ δυσκερή τεχνικά ζητήματα. Η ερευνητική κοινότητα είτε πρώτα για το ίτερ είτε για ό,τι έχει να κάνει με την πυρηνική σύνδεξη. Υπάρχει μεγάλη διάσταση, μεγάλος διχασμός και διαίρεση. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πρέπει να ληφθούν ε, δύσκολες πολιτικές αποφάσεις. Εδώ το θέμα είναι ότι πρέπει να ε, καταλάβουμε ότι μιλάμε για το ίτερ. Ανεξαρτήτως άλλων πολιτικών αποφάσεων που καλούμαστε να λάβουμε ή έχουμε λάβει κατά το παρελθόν. Ή προσπαθήσαμε να λάβουμε κατά το παρελθόν. Αυτή η συζήτηση όμως πρέπει να συνεχιστεί και με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο με παράδειγμα το ΙΤΕ και να εξηγήσουμε στα άλλα δύο θεσμικά όργανα ότι δεν μπορούν να ασκούν πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις στο Κοινοβούλιο λόγω των ε, διεθνών πιέσεων ή δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κομισιόν το Συμβούλιο. 6,6 εκατομμύρια μέχρι το 2020. Αναλαμβάνουμε αυτή τη δέσμευση και μετά η Δημοσιονομική Αρχή θα έχει το τελευταίο λόγο. Όταν υπήρξαν επίμαχα θέματα και κατά το παρελθόν, Υπήρξαν διαβεβαιώσεις κατέρωθεν συζητήσεις των επιτρόπων με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σχετικά με το μέχρι που μπορεί να φτάσει στις δηλώσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα, και αν θυμάμαι καλά, είχε δοθεί και η δυνατότητα να συμμετέχουν και ορισμένοι συγητές του Κοινοβουλίου στις συναντήσεις αυτές. Φαίνεται όμως ότι τα λησμόνησε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ITER. Ελπίζω στο μέλλον να διαμορφωθούν διαφορετικά, ώστε να μην βρισκόμαστε διαρκώς μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα. Ταυτόχρονα, στο τέλος της διαδικασίας, δεν θέλω να προκαταλάβω το τι θα συζητήσουμε ακόμη τις επόμενες εβδομάδες και το τι θα, ποιες αποφάσεις θα λάβουμε για το έργο αυτό που βεβαίως έχει μεγάλες διαστάσεις. Ο Καρλ Χάγκλουντ είπε επίσης ότι διεξάγεται συζήτηση και στην Επιτροπή Σούρε σε σχέση δηλαδή με συμβαστικές τροπολογίες για το λεγόμενο ring fencing ώστε να είναι ξεκάθαρη η χρηματοδότηση των έργων αυτών ταυτόχρονα μη στερώντας χρηματοδότηση από άλλα έργα. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι όταν προκύπτουν νέες ανάγκες εν τέλει πάντοτε υπάρχει συμμετοχή και από τα ε, πλαίσια από τα οποία προέρχονται τα έργα αυτά. Ωστόσο αυτό δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Κυρίως εν ώψη και των διαστάσεων του έργου αυτού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει με ηρεμία να σκεφτούμε αν μπορούμε να βρούμε άλλες ελκυστικές πηγές χρηματοδότησης και βεβαίως και για τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς των επόμενων μηνών. Όταν όμως προκαλείται τέτοια πίεση και αναμένονται κατεπηγόντως λύσεις, θα πρέπει να διευκρινιστεί πώς μέσα στην παρούσα κατάσταση αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις τους και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι και δωρητές για την χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ, ώστε να μην έχουμε μετά από λίγους μήνες εκπλήξεις και καλούμαστε να εξεύρουμε νέα χρηματοδότηση. Από ό,τι άκουσα, οι Ιάπωνες δήλωσαν ότι έχουν πρόβλημα μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα να παράσχουν τα όσα έχουν υποσχεθεί. Το 2008 νομίζω οι Ενωμένε Πολιτείες είχαν επίση βρεθεί σε δύσκολη ε, οικονομική θέση, το Κογκρέσο εν τω μεταξύ αποφάσισε να <clears throat> διακόψει τη συνεργασία με το έργο αυτό. Στο συνολικό, στη συνολική χρηματοδότηση δηλαδή δεν θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα και να καταλήξουμε σε ανώμαλη προσγείωση του χρόνου. Εάν δώσουμε πράσινο φως, γιατί το 2011 την δώσαμε, θα πρέπει αυτό να θυμόμαστε δηλαδή, και αν έχουμε εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση και μακροπρόθεσμα, ώστε να αρκέσει μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να πω ότι προσωπικά έχω εξασφαλίσει ότι η αντιπροσωπεία μας στο Κανταράσιο θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με την ανώτατη αρχή, διοικητική μάλλον αρχή, τον κύριο Μπερνάρ Μπιγκό που είναι υπεύθυνο ε, γενικός διευθυντής της ε, ε, Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και που είναι υπεύθυνο όσον αφορά τη Γαλλία για την παρακολούθηση του προγράμματος ITER. Είναι σε μόνιμη επαφή με τους Ιάπωνες και έχει μάλιστα συμβάλει, έχει στείλει και Γάλλους εμπειρογνώμους για να προσπαθήσει να βοηθήσει τους ε, Ιάπωνες να αρθμίσουν ε, το δύσκολο πρόβλημα της Φουκουσίμα και είναι επίσης υπεύθυνο αρμόδιος στη Γαλλία για το πρόγραμμα ενίσχυσης της σαρκοφάγου του Τσερνομπίλ. Οπότε θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά, αυτή τη φορά όλες τις ερωτήσεις που θα θέσει η αντιπροσωπεία μας, ίσως και νέες, ε, νέα ερωτήματα που, τα οποία απασχολούν την ίδια την Κομισιόν, ε, να μπορέσουν να λάβουν τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις σήμερα. Και από εκεί και μπρος ο εισηγητής μας θα μας κάνει προτάσεις. Κύριε θέλετε να κάνετε κάποιες τελικέ παρατηρήσει, πορίσματα, συμπεράσματα μάλλον. Πρόεδρε, πολύ καλή αρχική συζήτηση ήταν η κατά μου και παρακαλώ του συναδέλφου να τα στείλουν και γραπτό στα σχόλιά του. και φυσικά θα σας συντάξω εγώ ένα σχέδιο και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μεγάλη πλειοψηφία για αυτήν την υπόθεση γιατί είναι απαραίτητη δεδομένων των προκλήσεων που έχουμε από την διοικητική ε, άποψη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά και σας συγχαίρω γιατί στις εργασίες σας είστε μπροστά ε, σε σχέση με τις εργασίες της αρμόδιας επί Επιτροπής του Κοινοβουλίου που είναι η Επιτροπή Ήτρε η οποία δεν έχει ακόμα υιοθετήσει χρονοδιάγραμμα ούτε έχει ορίσει εισηγητή. Επί τη βάση των προβλέψεων λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε για τόσα γνωρίζουμε και από την εργασία στη ΣΥΤΡΕ, θα πρέπει να μπορούμε να τηρήσουμε το εξή χρονοδιάγραμμα. Πιο εις βάθος εξέταση του θέματος επί τη βάση ενό σχεδίου γνωμοδότηση στις 23 και 24 Μαου. Ίσως Εξέταση γραπτού, γραπτής έκθεσης της 16 ε, Ιουνίου, προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών ε, γύρω στις 16 Ιουνίου, να υιοθετήσουμε την έκθεση στην συνεδρίασή μας στις 12-13 Ιουλίου και έπειτα ψηφοφορία στην Ήτρε θα δούμε πότε θα γίνει για να δούμε και πότε θα περάσει από την Ολομέλεια η έκθεση αυτή. Προτείνω τώρα να επανέλθουμε στο σημείο 4 και 5 της ημερήσιας διάταξης. Σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 2011 επαριθμών 2. Όπως είχαμε ανακοινώσει στην προηγούμενη μας συνεδρίαση, βρισκόμαστε ενώπιον ενός ε, σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχει εκ νέου δυστυχώς να αποζημιώσει και να βοηθήσει κόσμο και χώρες που επλήγησαν από φυσικές από κλιματικές καταστροφές Σλοβενία, Κροατία και Τσεχία. Η συγκήτριά μας ε, Συνδόνια Γιουντρεύσκα δεν είναι εδώ. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Μπέγκη που είναι συνεισηγητής για αυτή την έκθεση. Για αυτές τις δύο εκθέσεις. Θα πω μόνο ότι μετά από τον τριμερή διάλογο που είχαμε με το Συμβούλιο υπό την ε, Ουγγρική Προεδρία και, και... κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήσαμε το σχέδιο διευθυντικού προϋπολογισμού υπαρθμών 1 και τον τρόπο χρηματοδότησης της βοήθειας στις ε, χώρες που επλήγησαν από πλημμύρες την περασμένη χρονιά μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία και η Πολωνία και όπου το Συμβούλιο είχε συμφωνήσει να ανατρέξει σε μια συνήθιστη διαδικασία αρνητικού αποθεματικού. Εμεί εκφράσαμε τι επιφυλάξει μας σε σχέση με αυτή την πρόταση και μάλιστα είχαμε πει πως αρνητικό αποθεματικό ήταν μια δυνατότητα περιορισμένη στα 200 εκατομμύρια ευρώ και ότι το σχέδιο διευθυντικού Προπολογισμού υπαριθμών 1 που ήδη είχε σχεδόν, εξαντλούσε σχεδόν ήδη το σύνολο αυτών των 200 εκατομμυρίων ευρώ και ότι εξάλλου η χρήση αυτής της διαδικασίας ε, δεν είχε ως αποτέλεσμα παρά το να αναβάλουμε για το τέλος του χρόνου μια επιλογή που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να γίνει όσον αφορά την ε, ίστατη χρηματοδότηση αν θα ήταν φρέσκο χρήμα ή αν θα ήταν ε, ανακύκλωση, αναδίπλωση και ανακατανομή των ποσών που ήδη υπήρχαν στον προϋπολογισμό. Δεν μπορέσαμε να πείσουμε το Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ δώσαμε πράσινο φως για την πρώτο διορθωτικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια, όπως το είχαμε προβλέψει και το είχαμε πει και στο Συμβούλιο, βρισκόμαστε τώρα ενώπιον του ίδιου προβλήματος με τις πλημμύρες που πάλι απαιτούν συνοδευτική βοήθεια και προσπάθεια από πλευράς του κοινοτικού προπολογισμού. Σλοβενία, Κροατία, Τσεχία. Η Κομισιόν πρότεινε φρέσκο χρήμα εδώ και το Συμβούλιο όμως δεν προσανατολίζεται προς αυτή τη λύση. Το Συμβούλιο θέλει να βρει πηγές ανακατανομής. Περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου για τις 23 Μαΐου και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να υιοθετήσουμε τη δική μας θέση αμέσως μετά. Το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε και για άλλους διορθωτικούς προπολογισμούς που είναι υπό προετοιμασία. Για την ώρα είναι μια ανταλλαγή απόψεων. Μπορούμε φυσικά να κάνουμε και από τη ουσία συζήτηση μετά από τις προτάσεις του εισηγητή μας σε επόμενη συνεδρίαση και με βάση τα όσα θα γνωρίζουμε για τη θέση του Συμβουλίου. Ο Ράιμερ, θες να μας πεις την άποψή σου, σε παρακαλώ. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπατε. Το υπαριθμόν 5 της ημερησίας ε, διατάξεως για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης μετά από τις πλημμύρες σε Σλοβενία, Κροατία και Δημοκρατία της Τσεχίας καταρχήν δεν παρουσιάζει προβλήματα. Μπορεί κανείς να δεχθεί και το ποσό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε βέβαια το αυξανόμενο πρόβλημα ότι το Συμβούλιο περιορίζεται σε συγκεκριμένες θέσεις του προϋπολογισμού 2011 χωρίς να λαμβάνει υπόψη απώλειες και με βάση την συζήτηση του τριμερούς διαλόγου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει ποια θέση θα λάβει. Αν θα δεχθεί την θέση του Συμβουλίου με το συνηθισμένο παιχνίδι, την συνηθισμένη αιτιολόγηση της ε, περιορισμένης απορρόφησης κονδυλίων ε, διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκαν επαρκώς ορισμένα κονδύλια, αν δηλαδή θα τα δεχθούμε όλα αυτά ή αν θα στηρίξουμε αυτά που προτείνει η συγγήτρια, δηλαδή πρόταση ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν λαμβάνει υπόψη περισσότερο, δεν διασυνδέει δηλαδή περισσότερο το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 3 με τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουμε τώρα. Αυτές τις πτυχές θα πρέπει να τις εξετάσουμε ξανά τις επόμενες εβδομάδες, 24, 24 Μαΐου. Μέχρι 26 Μαΐου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, μετά τον Ιούνιο ψηφοφορία στην Επιτροπή αυτά σε σχέση με τον προπολισμό, διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 3, σχετικά δηλαδή με τα ποσά, ώστε να δώσουμε ενδεχομένως ένα μήνυμα ή να αναζητηθούν άλλες λύσεις. Το ερώτημα αυτό τίθεται στις πολιτικές ομάδες. Κατά πόσον θέλουν να προχωρήσουν στην αντιπαράθεση αυτή, χωρίς ωστόσο η κινητοποίηση ή μη κινητοποίηση να οδηγήσει εν τέλει στην λήψη ομήρων των ε, χωρών μελών αυτών. Θα χρειαστεί λοιπόν θέση του Κοινοβουλίου η οποία να υποστηριχθεί βεβαίως από την απαραίτητη ε, ενισχυμένη πλειοψηφία. Δεν θα χρειαστεί να πω τίποτε περισσότερο ε, για την ώρα, αλλά όπως είπα θα πρέπει να ξανασκεφτούμε και εφόσον τώρα οι πρόσωποι εδώ του Συμβουλίου σημειώνουν τα όσα λέω, ίσως αυτό θα το δεχθούν και ως μήνυμα ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο όπως έχουν κάνει τις τελευταίες εβδομάδες, με κινητοποίηση δηλαδή ε, διορθωτικών προπολογισμών. Ευχαριστώ, ε, Ράιμερ. Δικαίως θυμήσατε το υπαριθμό 6 του, της, ε, μάλλον, της ημερησίας διατάξεως, σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 3. Ναι, είναι το συνηθισμένο βέβαια σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού που κλείνει τους λογαριασμούς του περασμένου έτους εξετάζοντας το δημοσιονομικό πλεόνασμα της διαχείρισης και προτείνοντας την επιστροφή του πλεονασμάτος αυτού στις χώρες μέλη. Το πλεονάσμα το οποίο ανέρχεται φέτος σε 4,5 ε, περίπου δισεκατομμύρια ευρώ ενώ το προηγούμενο χρόνο ήταν 2,5. Άρα υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, από χρόνο σε χρόνο. Τα 4,5 αυτά δις είναι πολλά. Εξηγούνται δε από την διαφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών. Για, κυρίως για την εμπορία αγροτικών προϊόντων. Για 185 ε, περίπου εκατομμύρια ευρώ. Τέλος πάντων, ένα, δις, δύο, 200 εκατομμύρια μάλλον, ε, είναι πια αυτά πραγματικός ίδιος πόρος και μάλιστα διαρκής. Και εξηγείται επίσης και από τη μη χρήση 2 δισεκατομμυρίων 700 εκατομμυρίων ευρώ πιστώσεων. Ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε διαμακρών την προηγούμενη χρονιά όταν ε, συζητούσαμε την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε υποβάλει τότε για μια τροποποίηση δηλαδή της δημοσιονομικής προοπτικής που να περιορίζεται βέβαια στην χρηματοδότηση του ε, προγράμματος ITER. Τα είχαμε συζητήσει αυτά βέβαια τότε, ε, ξανασυζητήσαμε σήμερα το πρωί. Έτσι εξηγούνται, έτσι κατανέμονται αυτά τα 4,5 δις πλεονάσματος. Και όπως είπε ο κύριος Μπέγκε, σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις μας θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια θέση αρχής. Θα προχωρήσουμε σε μια διασύνδεση εννοείται πολιτική μεταξύ των νέων αναγκών που εμφανίζονται κυρίως ε, στο ε, Ταμείο Αλληλεγγύης για το οποίο δεν υπάρχει για την ώρα διαθέσιμη χρηματοδότηση και σε αυτούς τους σημαντικούς πόρους που κανονικά θα πρέπει να επιστραφούν στις χώρες μέλη στα πλαίσια της διαχείρισης των υπολοιμάτων του 2010 ή θα δούμε τι θα μας προτείνει η Σιδονία, η συγκεντριά μας. Θα το σκεφτούν βεβαίως οι πολιτικές ομάδες, θα συνομιλήσουν και μεταξύ τους και η θέση του Συμβουλίου αναμένεται για τις 11 ή 14 έκτου και για λόγους διαδικαστικούς που έχουν σχέση με την διαβούλευση με τις Εθνικές Βουλές το χρονοδιάγραμμα θα είναι μάλλον σφιχτό για την ψήφιση αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 3. Αν δεν έχετε εσείς σχόλια, σας ευχαριστώ και προτείνω να περάσουμε στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεως Κοντά μας έχουμε τον Αντιπρόεδρο κύριο Καλφίν που τον ευχαριστώ για την έκθεσή του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ο οποίος προτίθεται να μας ενημερώσει για τον ανεπίσημο τριμερή διάλογο της 3ης Μαΐου. Έχετε το λόγο αγαπητέ φίλε. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε έναν εντατικό διάλογο με το Συμβούλιο στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Είχαμε στις 3 Μαΐου μία συνάντηση, έπεται μία ακόμη σήμερα το μεσημέρι και έχουμε προγραμματίσει μία τρίτη συνάντηση ε, στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε αυτό το τόσο ε, σφιχτό χρονοδιάγραμμα, γιατί θέλουμε, αν μπορούμε, μέχρι τα μέσα μένα να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Γιατί οι πληροφορίε που έχουμε από τι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου είναι ότι αυτή είναι η προθεσμία, αν θέλουμε να έχουμε αρκετό χρόνο για να κρίνουμε το τελικό κείμενο και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και μετά να δημοσιευθεί αυτό στην επίσημη εφημερίδα. για να μην υπάρξει ε, πρόβλημα και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ανησυχία. Ε, έχουν ε, υπάρξει αρκετά θέματα και εξελίξεις, θα ήθελα να σας ενημερώσω. Στην τελευταία συνεδρίαση της 3ης Μαΐου είχαμε δύο κείμενα τα οποία μας πρότεινε το Συμβούλιο. Το πρώτο θέμα αφορούσε τις οροφές τα ανώτατα όρια. Θα θυμάστε ότι είχαμε αποφασίσει αύξηση για όλες τις περιφέρειες και δι' για τη Μεσόγειο στο Κοινοβούλιο με βάση τις πολιτικές εξελίξεις ε, στη Βόρεια Αφρική. Αυτό είχαμε προτείνει ως Κοινοβούλιο. Η θέση του Συμβουλίου είναι ότι δέχονται αύξηση 4 δις ε, για την ε, Βόρεια Αφρική, όχι όμως για τις άλλες περιφέρειες. Επίσης, απορρίπτουν προς το παρόν την πρόταση να χρησιμοποιήσουμε 140 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε αυτή τη στιγμή για τη ναι, ε, Μεσόγειο και δεν θέλουν να συμπεριληφθεί ο συλλογισμός που έχουμε εμείς ε, προτείνει για να αιτιολογήσουμε την αύξηση αυτή και σε σχέση με την επιλεξιμότητα για άλλες χώρες. Είπαν ότι θα είμαστε υπέρ μόνο αν εστιάσουμε μόνο στη Βόρεια Αφρική και έχουμε αυτό την επιπλέον την αύξηση του ανώτατου ορίου. Και αν αυτό δεν ληφθεί στην επόμενη εντολή, στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, να είναι άπαξ δηλαδή αυτό το μέτρο. Αυτή είναι η θέση του Συμβουλίου. Επίσης, κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον σε σχέση με τα όσα προτείνει το Συμβούλιο, είναι να μπει αρχή της ε, conditionality, της αιρεσιμότητας. Να έχουμε δηλαδή μια πολιτική πρόοδο ρυθμίσει, Αυτή να είναι προπόθεση. Αυτό ακούγεται ωραίο, αλλά δημιουργεί κάποια πρακτικά προβλήματα. Και συγκεκριμένα, ποιο είναι αυτό που θα εκτιμήσει την πολιτική πρόοδο και τι ακριβώ συνιστά πολιτικό πρόοδο, πώ η τράπεζα θα γνωρίζει τι μπορεί να κάνει και ποια είναι τα όρια κτλ. Άρα, το θέμα των ανώτατων ορίων ακόμα είναι ανοιχτό. Λόγω των πρόσθετων κονδύνων που θέλουμε εμείς για άλλες περιφέρειες και δι για τις ε, χώρες που είναι σε προενταξιακή διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σχεδόν πρέπει να σταματήσει οι νέες επιχειρήσεις μέχρι το τέλος της ε, εντολής. Και το θέμα της ρεσιμότητας. Τι προτείνει το Συμβουλίο. Η Κομισιό να αποφασίσει για την αρεσιμότητα, για τις προϋποθέσεις και να δώσει το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Είπαμε ότι θα μπορούσαμε προκειμένου να δεχθούμε ενδεχομένω τη χρήση κατεξουσιοδότηση πράξεων. Δηλαδή να αποφασίζει μεν η Κομισιόν, αλλά να ενημερώνει το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο, και το Κοινοβούλιο να έχει τη δύναμη να σταματήσει την απόφαση, αν δεν τη θεωρήσει σκόπιμη. Αυτό είναι προσυζήτηση. Το δεύτερο τώρα. Και αυτό σχετίζεται με την αιρεσιμότητα. Υπάρχει μια πρόταση η οποία προήλθε από εμάς μετά από διαπραγματεύσεις επί του κειμένου για την εισαγωγή μιας, ε, ενός κριτηρίου ρεσιμότητας και σε ό,τι αφορά τις χώρες της εταιρική ε, σχέσης προς Ανατολάς. Δηλαδή να έχουμε την αρχή όσο περισσότερες μεταρρυθμίσεις τόσο περισσότερα κονδύλια θα είναι διαθέσιμα. More for more όπως λέμε. Αν καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο να βρούμε ένα μηχανισμό να εισαγάγουμε την αρχή της αρισμότητας. αυτό μπορούμε να το κάνουμε και για την νότια διάσταση και την ανατολική διάσταση. Και αυτό θα σηματοδοτήσει μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη βοήθεια και τη χρηματοδότηση από εδώ και πέρα. Γιατί ναι, μεν υπάρχει η αρεσιμότητα μέχρι να ληφθεί απόφαση, αλλά μετά υπάρχει ένα πράσινο φως, αυτόματα ρέουν τα κονδύλια από πολιτικής πλευράς ε, φαίνεται δελαστική η εισαγωγή της αρχής της αρισιμότητας, αλλά ίσως να μπορεί να είναι αποδεκτή και πάλι βέβαια μπορεί να δημιουργήσει ε, πρόσφορο έδαφος για αλλαγές στο μέλλον. Αλλά, όπως είπα, από τη στιγμή που μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για ένα μηχανισμό αξιολόγησης αυτής της αιρεσιμότητας και της αλλαγής χρήση των κονδυλίων. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα που συζητούμε αυτή τη στιγμή και υπάρχει και το δεύτερο ζήτημα των κατεξοδότηση πράξεων. Επιμένει πολύ σε αυτό το Κοινοβούλιο, είναι κατά η Κομισιόν και το Συμβούλιο, τι εννοούμε κατά εξοδότηση πράξη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλουμε να τι χρησιμοποιήσουμε για τι περιφερειακέ κατευθυντήριε γραμμέ. Η Κομισιόν και η Τράπεζα εκπονούν κατευθυντήριε γραμμέ για τι περιφέρειες, συγκεκριμένα ε, σε σχέση με το τι λέγεται στην εντολή, αλλά θα πρέπει να τι υποβάλουν στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και αν υπάρξει σιωπηρή συνένεση, προχωρούν. Εάν όχι, υπάρχει ε, πλέον η αναθεώρηση. Εμείς ε, βλέπουμε ότι η Κομισιόν, το Συμβούλιο και η Τράπεζα δεν θέλουν να μας δώσουν α, πολιτικά έγγραφα, περισσότερα πολιτικά έγγραφα. Εμείς πρέπει να βρούμε μια διέξοδο, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, τα είπαμε και χθε, για να δούμε πώς σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε και ίσως να καθορίσουμε κάποιες γενικές ε, προϋποθέσεις, γενικούς όρους, ένα χωριστό παράρτημα ε, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Και αυτό το παράρτημα ενδεχομένως θα μπορούσε στο μέλλον να αλλάξει με μια κατεξουσιοδότηση πράξη και έτσι να έχουν ε, το ελευθέρας για να δουν και να επεξεργαστούν τις συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένους όρους, που ίσως να μην θα ενδιαφέρει πολιτικά το Κοινοβούλιο τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν το δεύτερο. Πρώτο θέμα οροφές και αιρεσιμότητα και δεύτερο κατεξουσιοδότηση πράξης. Υπάρχει και ένα τρίτο, κάτι στο οποίο έχουμε επιμείνει πολύ. Η Λευκορωσία να μην είναι επιλέξιμη προς το παρόν και να μην υπάρχει υποσημείωση για την Ισλανδία. Άρα να θεωρείται υποψήφια χώρα Ισλανδία και να μην περιλαμβάνετε, να μην ενέχετε στα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν με τις κάτω χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο με τα συνταξιδοτικά κονδύλια. Αυτό που θέλει να κάνει το Συμβούλιο και προτείνει η Κομισιόν είναι η Ισλανδία να είναι ως επιλέξιμη χώρα μόνο αν λυθεί αυτό το ζήτημα. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα μέσα και έχουμε και υποθέσεις ε, ε, του δικαστηρίου. Θεωρούμε λίγο υπερβολικό λοιπόν αυτό που προτείνεται. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφωνία σε ό,τι αφορά την ε, Μεσογειακή Τράπεζα την Τράπεζα της Μεσογείου. Είναι πολύ αντίθετη η Κομισιόν πάνω σε αυτό. Και έχουμε και κάποια θέματα όχι τόσο σημαντικά, αλλά ε, ίσονο σημασία τέλο πάντων. Κάποιε ε, διαφορέ, διαφωνίε ό,τι αφορά τη διατύπωση, εστίαση μεγαλύτερη στην ανάπτυξη. Θέλουμε να λαμβάνονται υπόψη περισσότερο τα κριτήρια που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αξιολόγηση, δεν ικανοποιεί αυτό την τράπεζα. Τέλο πάντων, εμεί θέλουμε αυτό να συμπεριληφθεί στη διατύπωση. Και προ το παρόν κάτι τελευταίο. Το Συμβούλιο δεν στηρίζει, δεν είναι υπέρ τη ύπαρξη οποιοδήποτε μηχανισμού όπως προτείναμε σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια για το μέλλον και πώς θα πρέπει να οργανώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και διμερός και πολυμερός για την αναπτυξιακή βοήθεια στο μέλλον. Είναι ένα λεπτό ζήτημα πολιτικής πλευράς, απρόθυμο το Συμβούλιο, αλλά ανοιχτό το θέμα ακόμα. Δεν υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από πλευρά Συμβουλίου. Αν προβάλλουν στεναρή αντίσταση θα πρέπει να δούμε ποιε επιλογές έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό επειδή είναι σημαντικό. Και οι σοφοί έκαναν κάποιες πολύ σημαντικές συστάσεις στο έγγραφό τους. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν τη νέα εντολή και του χρόνου θα πρέπει να αρχίσει να βλέπει ε, την εντολή μετά το 2013 το Κοινοβούλιο και ίσως τότε θα είναι και πιο ξεκάθαρα αυτά τα βασικά θέματα. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι, ε, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αν το Συμβούλιο εργαστεί σκληρά μπορεί να κλείσει το θέμα μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αλλά εγώ έχω τις αμφιβολίες μου γιατί και αυτοί έχουν τις δικές τους διαδικασίες στο Συμβούλιο. Τα θέματα αυτά είναι θέματα για τα οποία διαφωνούμε ακόμα, αλλά από πλευράς μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ή άλλως. Και θα δούμε αν μπορούμε να υποχωρήσουμε σε κάποια θέματα ή όχι. Αλλά πολλά από τα κείμενα που έχουν εγκριθεί νομίζω ότι πρέπει να ε, θεωρήσουμε ότι ικανοποιούν το Κοινοβούλιο γιατί συμβαδίζουν με τις θέσεις μας. Ευχαριστώ. Euh, σα ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι, σα ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο δεξάγεται αυτέ τι διαπραγματεύσει. Βλέπουμε ότι για διάφορα σημεία υπάρχουν ακόμα ε, διαφορέ με το Συμβούλιο για σημαντικά θέματα. Και επίσης είναι θέμα το πρόβλημα μάλλον της ε, πολιτικής αιρεσιμότητας των δανείων ε, της ΕΤΕΠ ε, και επιπλέον της αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό το θέμα θα τεθεί με διαφορετικούς όρους μετά από τα γεγονότα στον αραβικό κόσμο. Μέχρι στιγμής για την πολιτική αιρεσιμότητα είχαμε εισάγει, στη, την είχα, εισάγει μάλλον στις συμφωνίες μας και σχεδόν ποτέ δεν την είχαμε λάβει υπόψη. Είναι σαφές όμως ότι είναι ρήτρε που είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν, αλλά που δεν θα μπορέσουμε πλέον από εδώ και στο εξή να αγνοήσουμε με τα όσα γίνονται στην άλλη όχθη της Μεσογείου. Δεν θα μπορούμε πια να χειριστούμε με τον ίδιο τρόπο τις χώρες που είναι σε πραγματική δημοκρατική μετάβαση και τις χώρες που με κάθε τρόπο προσπαθούν να την καθυστερήσουν. Πολύ συχνά δε η βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι στιγμής έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύσει αυταρχικά καθεστώτα στην εξουσία. Και σε ορισμένε ε, περιπτώσεις μάλιστα ε, χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι ενισχύσεις προς όφελος των εκάστοτε ε, αρμοδίων ηγετών. Αυτή είναι η φιλοσοφία λοιπόν και είναι πολύ σημαντικό θέμα και έχετε δίκιο που το φύγετε. Άρα λοιπόν, τι συνέχεια έχουμε, τι συνέχεια προβλέπετε, έχετε άλλη συνεδρίαση σήμερα κιόλας. Ωραία, θα μας πείτε λοιπόν τις εξελίξεις για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Αλλά είμαστε ευτυχείς πάντως που αυτό το σημαντικό θέμα βρίσκεται σε καλά χέρια. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, να σας ευχαριστήσω. Έχουμε εξαντλήσει την ημερήσια μας διάταξη. Η επόμενή μας συνεδρίαση είναι στις 23 Μαΐου στις 3. Ε, 23 και 24 Μαΐου κλείνω τη συνεδρίαση και κρατώ λίγα λεπτάκια τους συντονιστές. πέραστε συνεδρία σας λοιπόν και θα ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας σε τρία λεπτά.